everybody. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σε όλους. Ζητώ συγγνώμη που άργησα να ε, έρθω, αλλά πρέπει να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται τα ρολόγια στις διάφορες αίθουσες συνεδριάσεων δεν είναι συγχρονισμένα. Είχαμε μια συνεδρία τώρα το πρωί, ήταν εκεί η Ελίζα Φεράρα, το ρολόι έτυχε άλλη ώρα. Γι' αυτό αργήσαμε. Αλλά Ας, προχω... ξεκινήσουμε αμέσω. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει τη μητρική του. Έχουμε πλήρες γλωσσικό καθεστώς. Καθότι δεν έλαβα καμία πρόταση για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης, θεωρώ ότι εγκρίνεται, δεν έχουμε ανακοινώσει του Προέδρου. και έχετε λάβει και τα πρακτικά ε, των τελευταίων συνεδριάσεων. Σήμερα θα θέλαμε να συζητήσουμε, και είναι ουσιαστικά το μόνο μας θέμα, την έκθεση, την ενδιάμεση έκθεση, όπως την έχει υποβάλει η Υπερβάνσ. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Ξέρετε ότι η αρχική εκδοχή του κειμένου είναι η γαλλική, κατόπιν λάβαμε την αγγλική μετάφραση, τώρα όμως ε, έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Περβάνς. Η Περβάνς έρχεται. Είναι καθοδόν. <clears throat> Ότι μου ένα λεπτό να ολοκληρώσω και θα σου δώσω το λόγο. Ε, τη συζήτηση θα την εξής. Η εισηγήτρια θα ξεκινήσει τη συνεδρίαση, θα, μετά θα έχουμε ανοιχτή συζήτηση και η εισηγήτρια κατόπιν θα συνοψίσει. Νομίζω ότι θα έχουμε έντονη συζήτηση, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ότμαρ, έχει το λόγο. Η συγγήτρια ήρθε, αλλά κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας πω ότι στην ημερήσια διάταξη λέει απόφαση σχετικά με την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στο σημείο 4 της έκθεσης. Καθότι υπάρχει πια το κείμενο μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες από χθε, τουλάχιστον και τη δική μου πολιτική ομάδα, αλλά και για άλλες ε, πολιτικές ομάδες φαντάζομαι, έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Εάν θέλουμε να εμείνουμε στο στόχο, να έχουμε ευρία βάση υποστήριξη για την έκθεση αυτή, τότε το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση των τροπολογιών, 15 Ιουνίου δηλαδή, είναι υπερβολικά σύντομο χρονικό διάστημα. Την προηγούμενη εβδομάδα οι περισσότεροι από τους υπεύθυνου ήμασταν στην Κίνα. Την ε, Κυριακή στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, και δύο μέρες... Μάλλον θα έχουμε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες και δύο μέρες μετά στις 15 ε, Ιουνίου θα είναι η προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών. Στην πολιτική μου ομάδα είπα ότι θα πρέπει εντός της ομάδας μας να έχουμε κάποιο συντονισμό για να μπορούμε να συνοηθούμε με την εισηγήτρια. Θα παρακαλούσα λοιπόν να αλλάξουμε τη διαδικασία. Ε, αυτό θα διευκολύνει και την εξέβρεση συνένεσης. Θα παρακαλούσα λοιπόν την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών να τη μεταφέρουμε κατά μία εβδομάδα, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα εσωτερικά αλλά και με την εισηγήτρια να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε πριν την κατάσταση των Η 15 15η μου φαίνεται πολύ σύντομη προθεσμία. Ο Τμάρ, για το σημείο αυτό ήθελα... Το σημείο αυτό ήθελα να το συζητήσω μετά την συζήτηση της έκθεσης. Ε, σήμερα το απόγευμα έχουμε και την συζήτηση με το πάνελ των εμπειρογνωμόνων, με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω και στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε μία έκθεση την οποία να στηρίζει αν όχι κάθε βουλευτή το τουλάχιστον μια σημαντική πλειοψηφία. Δεν θέλουμε λοιπόν να στηριζει αν οχι καθε βουλευτη στο τουλαχιστον μια έκθεση η οποία να μην βρει την υποστήριξη της ε, πλειοψηφίας. Ε, γι' αυτό, Ότμαρ, συμφωνώ με την εκτίμησή σου. Πράγματι, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα επιστρέψουμε από την Αμερική και δύο μέρες μετά είναι η λήξη της προθεσμίας. Είναι πολύ λίγος χρόνος αυτός. Ε, μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα το θέμα αυτό. Ε, κατάλα... θα το είχα συζητήσει το θέμα αυτό στο τέλος της συνεδρίας, αλλά τέλος πάντων. Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα Άλτε συζήτησε το ίδιο θέμα και έχει τα ίδια προβλήματα. Συμφωνούμε λοιπόν με αναβολή για την κατάσταση των τροπολογιών κατά μία εβδομάδα ή κάτι τέτοιο. Διότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες σχετικά με την έκθεση αυτή και πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο να καταλήξουμε σε συνένεση εάν Έχουμε περισσότερο χρόνο. Συμφωνούμε λοιπόν με αυτό που είπε ο Ότμαρ Καράς. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Γκίγκολτ. Ναι, συμφωνώ με τις ανησυχίες αυτές. Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο για να διευκολύνουμε την ε, εξέβριση συμβιβασμού, όχι μόνο να δώσουμε μια εβδομάδα παραπάνω για συνεδρίαση εντό των ομάδων, αλλά να την εκμεταλλευτούμε την εβδομάδα αυτή και για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στι ομάδες όπως γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις ε, συμβιβασμού, για να έχουμε μια αίσθηση για το ποιε είναι οι ανησυχίε των άλλων στην όλη διαδικασία αυτή, διότι αλλιώ μπορεί να μην κερδίσουμε και πολλά με την επιπλέον εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ε, χρησιμοποιήσουμε το χρόνο αυτόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Άλβαρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω γιατί όπω είπε ο Ότμαρ, η ισπανική μετάφραση δεν υπάρχει. Και ε, Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ βραχυπρόθεσμη η ημερομηνία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο για να έχουμε και τις μεταφράσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. I fully support Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα είναι χρήσιμη μια παράταση. Προσπαθήσαμε να ε, συνοηθούμε με τους ε, συναδέρφους μας ε, και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να συντονιστούμε. Φαντάζομαι ότι οι μεγαλύτερε πολιτικέ ομάδε θα έχουν ακόμα μεγαλύτερε δυσκολίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νότμαρ Καράς όχι μόνο για την πρότασή του, αλλά και το περιεχόμενό της και το πνεύμα υπό το οποίο την έκανε. Ίσως είναι μια ε, υπερβολική ταπεινοφροσύνη εκ μέρους μου, αλλά θα ήθελα να γίνει μια συζήτηση με όλες τις πολιτικές ομάδες. Και αν θέλουμε να υπάρξει μια καλή συζήτηση, θα πρέπει στο εσωτερικό της πολιτικής ομάδας να, γίνει, να οργανωθεί μια σωστή δουλειά συντονισμού πάνω σε μια καλή βάση γιατί αλλιώς υπάρχουν απογοητεύσεις, ε, κατατίθενται κάποιες ε, τροπολογίες από που δεν έχουν συζητηθεί. Οτιδήποτε επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ενισχύσει τη γραμμή του είναι ευπρόσδεκτο. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω ότι το κατευθυντήριο νήμα της έκθεσης που είναι η βάση των διαπραγματεύσεων ε, νομίζω ότι δεν παρουσιάζει δυσκολίες. Θα πρέπει μόνο να αναλύσουμε κάτω από ποιες ε, προϋποθέσεις ή τις ε, διολυστήσεις συνεπάγεται σε σχέση με την Ολομέλεια και την ψηφοφορία εκεί, καθώς και στην Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι ο στόχος να έχουμε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή πριν από το καλοκαίρι θα πρέπει να παραμείνει βασικός μας στόχος γιατί αλλιώς ε, αν δούμε τι γίνεται εκτός του σώματος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για παράδειγμα, η δύναμη του δικού μας μηνύματος θα αμβλυνθεί. και νομίζω ότι κανένα μέλος αυτής της Επιτροπής δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν δυσκολίε επί της βασικής αρχής. Και θα ήθελα να πω σε όλες τις πολιτικές ομάδες τη διαθεσιμότητά μου και για να συναντηθώ με εκείνους που επιθυμούν να διευκρινίσουν κάποια πτυχή της έκθεσης πριν από τη σύνταξη των τροπολογιών και πριν από τη διαπραγμάτευση των συμβαστικών τροπολογιών. Εάν θέλουμε να ψηφίσουμε, όπως είπες, ε, Περβάνσο, στην Επιτροπή πριν από τη θερινή πάυση, ποια θα ήταν η τελευταία δυνατότητα. Πότε θα ήταν η τελευταία δυνατότητα να διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να, έχουμε, να, να συγκληθεί μια έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής. Το ερώτημά μου είναι ο πρόεδρος λέει το εξή. Ο κύριος Γκέτς μου έδειξε το μέγιστο διάστημα που θα μπορούσαμε να ορίσουμε σε σχέση με την ε, προθεσμία εκπνοής των τροπολογιών. Δηλαδή 22 Ιουνίου. Δεν είμαι βέβαιος ότι μια εβδομάδα είναι αρκετή, εάν πράγματι θέλετε να γίνει αυτή η δουλειά. Μία εβδομάδα είναι εντάξει για όλους. Το δέχεστε. Άρα 22 ή 23 Ιουνίου κύριε Γκέτς. Τι λέτε. Αν λέμε μία εβδομάδα είναι 22 Ιουνίου. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να πάμε ως τις 23. Ξέρουμε πότε είναι μία εβδομάδα. Οι μεταφράσεις θα μπορούσαν να είναι πρόβλημα, αλλά αν έχουμε την μετάφραση σε κάποιες γλώσσες κλειδί, ε, αυτό θα πρέπει να μας αρκεί. Συμφωνούμε λοιπόν τώρα, ομόφωνη απόφαση ότι θα παρατείνουμε την προθεσμία την κατάθεση τροπολογιών κατά μία εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Εντάξει, ωραία. Μεσημέρι, 12 η ώρα. Αυτά λοιπόν. Περνάμε τώρα στο θέμα της σημερινής συζήτησης και θέλω να καλέσω την Περβάνς να παρουσιάσει και πάλι κάποια σημεία κλειδιά για κατόπιν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα που όλοι είχατε την δυνατότητα να διαβάσετε την έκθεση στη μητρική σα γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ήδη προηγήθηκε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στι 17, στις 18 Μαΐου, λέει ο μιλήτρια στο Στρασβούργο, ε, και τότε λίγα μόνο μέλη είχαν μπορέσει να ασχοληθούν ε, με, το, με την έκθεση και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η σύνταξη αυτή τη έκθεση είχε ολοκληρωθεί στι 6 Μαου και ότι έκτοτε πολλά πράγματα συνέβησαν τα οποία προφανώς ε, εκείνη την εποχή δεν αναφέρονται στην έκθεση αλλά θα αποτελέσουν ε, το αντικείμενο συζήτησης όταν, σε σχέση με τις τροπολογίες που θα υποβληθούν. Στην ανάλυση που επιθυμώ να προτείνω εν σχέση με τα όσα συνέβησαν μετά την 6η Μαΐου, είναι και η νέα αξιολόγηση που δόθηκε στη νέα διάσταση της κρίσης. Και επιθυμώ, ανοίγοντας τη σύντηση σήμερα, να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί νομίζω ότι συμφωνεί με το πνεύμα της έκθεσης, έτσι όπως το έχετε στα χέρια σας σήμερα. Πολλοί αναλύουν τη νέα εξέλιξη της κρίσης ως ε, κρίση του εθνικού χρέους. Νομίζω ότι το να προσδιορίζει κανείς την κρίση σε συνάρτηση, ως κρίση μάλλον του εθνικού χρέους, είναι misleading, είναι παραπλανητικό, λέει στα αγγλικά η ομιλήτρια, για τις προτάσεις όσον αφορά την έξοδο από την κρίση. Γιατί αν υπάρχει μια κρίση εθνικού χρέους σε κάποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ένα διακύβευμα ε, γύρω από αυτό το εθνικό χρέος, το δημόσιο χρέος. Γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες που έχουν υπερβολικά χρέη και που δεν γίνονται αντικείμενο, αντικείμενο επιθέσεις από τις αγορές οι ελλείψεις που αναγνωρίζουμε εμείς στην έκθεση όσον αφορά τη λειτουργία υπό για κυβέρνηση Ευρωζώνης, της ανισορροπίας μεταξύ του νομισματικού και οικονομικού πυλώνα που θα πρέπει να εξεταστούν εκ του σύνεγγης ως στοιχεία του πλαισίου ε, για την ανάλυση αυτής της νέας διάστασης της κρίσης. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την έκθεση, έχουν γίνει πολλές προτάσεις και υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάλυσης μιας διάγνωσης την οποία ήδη παρουσίασα τελευταία φορά και δεν θα ήθελα να επανέλθω θα ήθελα απλώς να επισημάνω για τους συναδέλφους ορισμένες ε, παραγράφους που μου φαίνονται απολύτως ε, κρίσιμες στην έκθεση. Όχι επειδή θεωρώ ότι η θα πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα σημεία αυτά, αλλά θεωρώ ότι για μένα εκφράζουν τις ε, απολύτως ουσιαστικές, απαραίτητες ε, προτάσεις. Και θα διαβάσω αυτό τον ε, κατάλογο, γιατί νομίζω σε αυτό το στάδιο συζήτηση που έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι σημαντικό. Πρόκειται για την αιτιολογική σκέψη F, παράγραφο 20, 116, 122, 130, 133, 154, 168, 69 και 216. Γιατί λοιπόν επισημαίνω αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Γιατί είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία μας επιτρέπουν στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, έχω την άποψη, να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία οδό εξόδου από την κρίση και επιτρέπουν, εάν εφόσον συμφωνεί το Κοινοβούλιο, να περάσουμε το μήνυμα που θεωρώ ότι αναμένουν από εμά οι συμπολίτε μα, δηλαδή ένα μήνυμα ελπίδα. Ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πράξει κάτι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαθέτει ένα χρήσιμο επίπεδο παρέμβασης, όπου ούτω ώστε μεθαύριο ε, όπου βλέπουμε τι γίνεται στις ΗΠΑ ή στην Κίνα, πέρα από τις δυσκολίες της κάθε χώρας μέλος να αντιμετωπίσει την κρίση, ε, υπάρχει μια προσφορά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι φέρελπης υπό την έννοια της αύξησης τη αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας. Αυτό είναι το πνεύμα των προτάσεων που υποβάλλω. Δεν θα ήθελα να επισέλθω στι λεπτομέρειες, βασίζοντας στη διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες που δεν ασκεί επαρκώς και είναι μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες που τις έχουν εμπιστευθεί οι συνθήκες και να ε, ε, μιλήσει με μια ισχυρή φωνή γιατί έχει τα χρηματοπιστωτικά μέσα και όχι μόνον για να εφαρμόσει αυτές τις αρμοδιότητες ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος, προκλήσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να αναγνωρίσει πλήρως το Μάρτιο του 2007 όταν όρισε τη στρατηγική που ορισμένοι ονομάζουν ε, τέσσερις φορές 2020 μια στρατηγική βιωσιμότητα στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό τομέα και που δεν μπόρεσε να αναχιστεί μέσω αυτή τη κρίση. Ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω γιατί είναι σημαντικό στο πλαίσιο ανάλυση τη κρίση είναι η ισορροπία των προτάσεων που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι επί των οποίων οι G20 έχουν ενίοτε μια καποσφαιρική προσέγγιση η οποία επιτρέπει να εξετάσουμε την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων προτάσεων αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει πράγματι προτάσεις έτσι όπως καλούμε θα το πράξουμε στο στερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η δική μου ανησυχία ότι εξετάζουμε αυτές τις προτάσεις όσον αφορά την μεταρρύθμιση του κανονισμού των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών αλλά και τις εποπτείας από την άποψη της αποτελεσματικότητας, από την άποψη του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος, κοινής ευρωπαϊκής ωφέλειας, δηλαδή της μακροπρόθεσμης επένδυσης, χρηματοδότηση των επενδύσεων και των καινοτομιών, ούτε ώστε να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας ε, καθαρός ε, ε, εισφορέας σε σχέση με αυτό που αναμένουν οι πολίτες. Δηλαδή την επάνωδο σε ένα επίπεδο απασχόλησης για τον καθένα. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω η παρουσίασή μου είναι πολύ πλατιά, αλλά νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν την ευκαιρία από τις 18 Μαΐου, είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν διάφορες ε, προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση και είναι ακριβώς ιδίω αυτό το μήνυμα ελπίδας που πιστεύω ότι θα πρέπει να κομίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα αυτής της έκθεσης και που θα ήθελα ακριβώς ε, να αναφέρω σήμερα, χωρίς να επισέλθω στις λεπτομέρειες που θα τεθούν στο πλαίσιο της συζήτησης. Πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο, διαβάζω τα ονόματα. Πέτη Κάνεν, ε, Μπογκέζιο, Ντεγιόν, Τόμας Μαν και Μαντλένα Άλβαρες. Όλε Σμιτ, ο Πασκάλ, ο Τσμαρκάρας. Και πριν μπούμε στον δεύτερο γύρο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν που επίσης το ζήτησε. Ε, σχεδόν όλοι ζήτησαν το λόγο. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Thank you, Mr. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που λάβατε υπόψη σας την ανάγκη για περισσότερο χρόνο εργασίας πάνω στην έκθεση, διότι βασικός μας στόχος σε όλες τις πολιτικές ομάδες είναι να καταλήξουμε σε όσο γίνεται καλύτερη έκθεση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με βάση ε, την ε, ομοφωνία, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε την ε, πολιτική μόχλευση που θέλουμε για τις νομοδοτήσεις μας. Μ, πάρα, αρέσει πάρα πολύ η πολιτική. Μ' αρέσει που έχουμε διαφορετικές απόψεις ε, και διαφορετική ιδεολογική ερμηνεία. Αλλά ίσως να ερμηνεύουμε τις περιγραφές αυτές με κάπως διαφορετικούς τρόπους. Ε, νομίζω ότι αντικατοπτρίζουμε μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν ε, των ε, σοσιαλδημοκρατών. και έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το, το ποιο ήταν το λάθος στην νομοθετική ρύθμιση που οδήγησε στην παρούσα κατάσταση. Γι' αυτό θα ήθελα να αλλάξει η διατύπωση στην έκθεση ώστε να διαγράψουμε τους ε, ιδεολογικούς όρους και τις σχετικές περιγραφές. Όσον αφορά την κατάσταση και την Ελλάδα, υπήρχε νομοθετική ρύθμιση για το συγκεκριμένο θέμα και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο αγωνίστηκαν για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Φτάνουμε πάλι στο θέμα των κυρίαρχων κρατών. Τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο δεν θέλησαν να ακολουθήσουν τη γραμμή αυτή. Και θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της Ελλάδας, ε, ε, την οικονομική κρίση, την ε, δημοσιονομική κρίση και τις επιπτώσεις ε, στην ε, γενικότερη οικονομία. Μετά το θέμα της Ελλάδας, νομίζω ότι καλό θα είναι να τονίσουμε περισσότερο την ανάγκη για περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς τα κυρίαρχα κράτη προσπαθούν να χειριστούν τέτοιες περιπτώσεις ε, με τρόπο περιφερειακό τη στιγμή που τα προβλήματα είναι ε, παγκόσμια. Ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία με την εισηγήτρια για να μπορέσουμε να βρούμε μια συνεκτική προσέγγιση. Θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες ε, και πέρα από τα θέματα που έθιξα θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να τονίσουμε την προοπτική για ανάπτυξη, τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, της ε, κοινοπραξίας δημοσίου, δικαίου, ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη χρηματοδότηση και θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική διάσταση, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ένωση και την λειτουργία, τη λειτουργικότητα της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να αναπτύξουμε στα πλαίσια μιας καλής συνεργασίας. Στα επόμενα βήματα θα πρέπει να εξετάσουμε την ε, περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σαφές ότι αυτό θα πρέπει να είναι η βάση των ε, σχετικών προτάσεων. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην νομοθετική ρύθμιση. Ε, δεν αρκεί η νομοθεσία που έχουμε αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πορκέζια. Ο κύριος Πορκέζιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γενικά, Είμαι επικριτικός απέναντι στην έκθεση της κυρίας ε, Περές, παρότι υπάρχουν πολλά σημεία που συζητάνε πολύ σημαντικά θέματα με σωστό τρόπο. Η γενική μου εκτίμηση όμως είναι ότι η έκθεση αυτή είναι υπερβολικά πολιτική αν θέλετε. Και αυτό πρέπει να το επικρίνουμε. Ιδιαίτερα επειδή προτείνονται οικονομικές λύσεις χωρίς να δίδονται ακριβείς ε, πληροφορίες σχετικά με την πραγματική οικονομική πολιτική που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να βρουν μια στρατηγική εξόδου από την ε, οικονομική κρίση. Επίσης πιστεύω ότι μια τέτοια σημαντική έκθεση που είναι και η πρώτη της Επιτροπής μας θα πρέπει να ε, υποδεικνύει τους υπεύθυνους. Η κρίση που συζητάμε δεν εμφανίστηκε εν μία νυχτή από το τίποτα. Υπήρχαν αιτίε, υπάρχουν ευθύνε. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο ευρία οπτική της κρίσης. Πρέπει να καταλάβουμε από πού προήλθε και πού θα μας πάει. Θα κάνω και άλλες σχετικές παρατηρήσεις, για παράδειγμα. Θα ήθελα να σχολιάσω το σημείο 153, η πρόταση της Περβάνς για μια επιτροπή των σοφών, ωραία, πολύ καλά, στην οποία ε, να προεδρεύει ο Χέρμαν Φαν Ρόμπαϊ, εντάξει, ε, που θα είναι υπεύθυνη για την οικονομική διακυβέρνηση. Ο κύριος Φαν Ρόμπαϊ θα συμμετέχει επίσημα στην ε, συνάντηση της Ισπανίας της Λέσης Πίλτεπερκ και Θέλουμε η οικονομική κυβέρνηση να βρίσκεται στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και νομίζω ότι αυτό συνδέεται με τις αιτίες της οικονομικής κρίσης. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνονται λύσεις οι οποίες να μην προέρχονται απαραίτητα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που οδήγησαν στην κρίση στην πρώτη φάση. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Όσον αφορά συγκεκριμένε παρατηρήσεις, είμαι κατά της εισαγωγής νέων ευρωπαϊκών φόρων. Έχουμε πολλούς φόρους ούτως ή άλλως στις οικονομίες μας. Ε, νομίζω ότι αυτό θα στείλει λάθος μήνυμα στην πραγματική οικονομία αν ξεκινήσουμε μια τέτοια στρατηγική. Αυτό και εξαιτία τη σημασία ε, η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να δοθεί για την όθηση που πρέπει να δοθεί για το μεγάλο σύστημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε είναι γεωργικές είτε είναι βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ε, το κεφάλαιο 153 νομίζω, το οποίο αφορά ακριβώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι ουσιαστικά κάτι περιθωριακό, ενώ θα έπρεπε να είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Πρέπει να εξετάσουμε εις βάθος ποια είναι τα αίτια της ε, έλλειψης ε, ροής πιστώσεων στο σύστημα των μικρομεσαίων επιχειρώσεων. Ακόμα και όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έκανε και κάνει αυτούς τους μήνες συνδράμει το τραπεζικό σύστημα, υπάρχει ένα τεράστιο ποσό κεφαλαίων το οποίο εισραίει στις τράπεζες αλλά δεν φτάνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν φορολογικές πολιτικές αλλά και άλλες οι οποίες πολλές φορές ε, γονατίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ έχω και άμεση εμπειρία του θέματος αυτού στη χώρα μου. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στη λανθασμένη άγουσα κατ' εμέ, διότι δεν ε, θέτουμε στο ε, επίκεντρο της πολιτικής οικονομικής εξυγίασης το σύστημα αυτό. Όσον αφορά δε τον τραπεζικό κόσμο, είμαστε σε αντίστοιχη κατάσταση. θέλουμε ή δεν θέλουμε να λάβουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο που πρέπει να διεξάγουν τα συστήματα των ε, ε λαϊκών τραπεζών, των τραπεζών ε, που βρίσκονται επί τόπου. Επειδή ακριβώς πρέπει να είμαστε μια Ευρώπη των περιφερειών, νομίζω ότι αυτό λείπει στην έκθεση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να είναι ένα απόσπαστο τμήμα των πολύ χρήσιμων προτάσεων τις οποίες θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε. Για να περάσω τώρα στα αίτια και πάλι. Και τα μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθούν τα εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν στον οικονομικό κόσμο. Καταρχάς χρειαζόμαστε σαφείς και συγκεκριμένες διατάξεις ώστε ε, να ε, μην επιτρέπουμε στις τράπεζες να εκδίδουν ε, δομημένα προγράμματα. Στο City υπάρχει μια πολύ ε, ε, συγκεκριμένη έκφραση που αναφέρεται στο συνικό τείχος. Νομίζω ότι αυτό που έγινε για τον ασφαλιστικό τομέα στη χώρα μου θα πρέπει ε, να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να υψώσουμε αυτό το συνικό τείχος το οποίο θα περιλαμβάνει όλους αυτούς που εμπλέκονται στην κατάσταση. Ε, προέκυψαν ε, μεγάλες συγκρούσεις συμφερόντων στα πλαίσια αυτής της κρίσεως και ε, ελοχεύει ο κίνδυνο να μείνουν όσοι έχουν αυτά τα πράγματα εάν δεν τα λύσουμε. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ σοβαρό και θα ήταν δική μας ευθύνη, διότι δεν θα έχουμε εργαστεί αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση. E Χρειαζόμαστε μέτρα λοιπόν ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις ε, συμφερόντων ε, οι οποίες προκύπτουν και από τους οίκους αξιολόγησης. Οι οίκοι αξιολόγησης κανονικά θα έπρεπε να αξιολογούν μόνο τις κεντρικές τράπεζες και οι υπόλοιπες τράπεζες να είναι ανεξάρτητες της πολιτική ηγεσία και να μην αποτελούν αντικείμενο ε, διαπραγμάτευσης και εκβιασμού μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Ολοκληρώνω εντάχει να επισημάνω ότι στο θέμα των, ε, ε, της σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε οίκους ε, που έχουν ε, συμβούλους που κάνουν ε, και χρέη, τελούν και χρέη συμβούλου στις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος και οι ελεγχόμενοι και οι ελεγκτές τελικά είναι τα ίδια άτομα. Κάτι τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Ε, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη στην Πράσινη Βίβλο ε, και να πω εδώ ότι ο υπουργό ε, Μαρόνι στην Ιταλία το εισήγαγε και θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη στρατηγική η κρίση θα μας επιτρέψει να συμπεριλάβουμε στο ευρωπαϊκό μοντέλο, συμπληρώνοντας την κοινωνική και οικονομική μας κουλτούρα, το γεγονός ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια οι εργαζόμενοι, να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Δεόν. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να συγχαρώ την κυρία Περβάνς για το έργο της. Οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται αυτή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία έκθεση η οποία έχει λάβει τα κοινωνικά θέματα υπόψη. Και νομίζω ότι αυτό σίγουρα μπορούμε να το πούμε σε αυτή την περίπτωση. Θα προτείνουμε σίγουρα κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά ε, με ενδιαφέρουν κυρίως δύο πράγματα. Καταρχάς η ανάλυση. Ε, έχουμε στη διάθεσή μας περιορισμένο αριθμό σελίδων, αυτό είναι αλήθεια, αλλά για τον μέσο πολίτη είναι πολύ δύσκολο να διαβάσει αυτή την τόσο τεχνική ανάλυση. Και ναι, μεν θα πρέπει να υπάρχουν τα τεχνικά στοιχεία, διότι πρέπει να επιλύσουμε τεχνικά προβλήματα, αλλά στην εισαγωγή της έκθεσης ίσως θα έπρεπε να αναφερόμαστε λίγο περισσότερο σε αυτή την οτροπία η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αναφέρομαι σε αυτή την ε, ε, νοοτροπία εμπιστοσύνη στην αγορά. Υπάρχουν πραγματικοί επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν κινδύνους, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία ε, κερδοσκοπία και μία απόπειρα να γίνει ο καθένας ε, πλούσιος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και επομένως ε, θέτουμε έμφαση αποκλειστικά και μόνο στην αγορά και ξεχνούμε όλα τα υπόλοιπα. ναι μεν υπήρχε μια εξωτερική εξέλιξη, αλλά τα κράτη-μέλη συνειδητά επέλεξαν μια, να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η κρίση αυτή μας έμαθε κάτι, μας ε, έμαθε την κερδοσκοπία, ε, και όλα αυτά προέκυψαν από την ε, τεράστια εμπιστοσύνη στην αγορά και στην πεποίθηση ότι μπορεί να λύσει τα πάντα. Λείπει ένα στοιχείο από την έκθεση. Ο τίτλος είναι πάρα πολύ μεγάλος, η χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση και επομένως δεν θα πρέπει να περιοριστούμε απλά και μόνο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και ανησυχώ όταν διαπιστώνω ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ χρειάστηκε να λάβει ε, κρατική επιδότηση και υποστήριξη για όλες τις ε, αυτοκινητοβιομηχανίες. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο τραπεζικό τομέα. Αυτό συμβαίνει και στην πραγματική οικονομία, διότι θα πρέπει να εξεύρουμε λύσεις. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες για να αποτύχουν, too big to fail. Τίθεται το ερώτημα, της συνεισφοράς του πολίτη, του φορολογούμενου για την ε, ε, διάσωσή τους. Το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρεται σε λύσεις από ευρωπαϊκής πλευράς ε, είναι κάτι το οποίο είναι θετικό. Αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα. Αν δούμε όλα αυτά τα οποία πρότεινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρονται σε μια προσαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, και Ανάπτυξης και οι δράσεις είναι λιγότερες ως προς την ε, καταπολέμηση της ε, ένδυας, τόσο όσον αφορά τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Ε, πολύ μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών ζουν κάτω από το όριο της φτώχεια. φτώχειας και επομένως οι περικοπές οι οποίες πρέπει να γίνουν ε, σημαίνουν ότι θα μειωθούν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Αφενός λοιπόν έχουμε τις περικοπές και αφετέρου έχουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο θα πρέπει να παραμείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Η Ευρώπη δεν κατάφερε να βρει μια ισορροπία στο θέμα αυτό. Γι' αυτό απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση στην Ευρώπη. Η ε, έδωσε έμφαση στα κοινωνικά στοιχεία, αλλά ε, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα κλίμα εμπιστοσύνης για τα θεσμικά όργανα από τα οποία ζητούμε να εξεύρουν τις λύσεις. Ε, υπάρχουν και κάποιες ε, ανθυπολεπτομέρειες, δεν θα τις συζητήσω εδώ. Το θέμα της διακυβέρνησης και η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις έγινε μια έρευνα από την οποία προκύπτει ότι η πλειονότητα των Ολλανδών είναι υπέρ της ε, συμμετοχής των εργαζομένων ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας ε, επιχείρησης. Μάλιστα μιλούν για το ίμιση των μελών. Θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένε προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όλα αυτά τα θέματα είναι ίσιον σημασία και δεν θα επιμείνω σε αυτά. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Μαγδαλένα. Η Μαγδαλένα Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε τη σημασία αυτού του κειμένου και νομίζω ότι η Περβάνς πραγματικά έκανε μια θαυμάσια εργασία από την άποψη της ανάλυσης των αιτιών της κρίσης, των επιπτώσεων και αυτό οδήγησε μια σειρά μέτρων. Συμμερίζομαι την άποψη ότι το πρώτο στο μέλημά μας είναι να προστατεύσουμε τον πολίτη και αυτή η προστασία συνεπάγεται μια ενίσχυση των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η Ευρώπη για να το επιτελέσει αυτό το έργο. Ούτως ώστε να λάβει μέτρα τα οποία ενισχύουν αυτές τις δυνατότητες. Νομίζω ότι σε αυτό το κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε στη γραμμή της πρωτοπορίας, να επιφέρουμε αλλαγές και να φέρουμε στο τραπέζι νέες ιδέες. Νέες ε, ιδέες που τις βλέπουμε και σε αυτή την ε, έκθεση σε σχέση με, την, ε, με τους, ε, για παράδειγμα με την ανάλυση των οίκων, του ρόλου των οίκων πιστοληπτικής, αξιολόγηση των οίκων αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Τώρα, όσον αφορά το Σύμφωνο ανάπτυξη και Σταθερότητας, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, δυνατότητα ανάπτυξη τη Ευρώπης και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Συνεπώς, θα πρέπει να ερμηνεύσουμε το Σύμφωνο ανάπτυξη και σταθερότητα, δίδοντα δυνατότητε στην ε, χρηματοπιστωτική παγιοποίηση ώστε να λάβουμε μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων που να μας επιτρέπουν διαρθρωτικές αλλαγές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Ε, Αυτό είναι το σημείο στο οποίο θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη εμβάθυνση στο κείμενο ούτως ώστε να ερμηνευθεί υπό τη σωστή έννοια το σύμφωνο σταθερότητας που θεωρώ ότι εμφανίζει κάποιες ανισορροπίες όσον αφορά μόνο την, ε, όταν αφαίρεται αποκλειστικά και μόνο στην ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις επενδύσεις και ποια είναι επίσης, ποιοι είναι οι δείκτες της εκπλήρωσης αυτής της συνθήκης. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Ο Τόμας Μάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήδη στην πρώτη παρουσίαση της έκθεσης της Περβάνσα ε, μπόρεσα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι στο να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια συντομότερη εκδοχή αργότερα, θα πρέπει να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες. Και συμφωνώ ότι η έκθεση δεν θα πρέπει να έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Αυτό θα πρέπει να μπορούμε να το κατορθώσουμε. Και ε, νομίζω ότι έχουμε μια καλή ευκαιρία να δει το φως στο τέλος ένα έγγραφο αρκετά ισορροπημένο θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να λέμε, νομίζω ότι είναι σωστό να, έχουμε, να θέσουμε κάποια κριτήρια στη μελλοντική ανάπτυξη και μεγέθυνση να δούμε τι σημαίνει ποιοτική ανάπτυξη. Γιατί χρειαζόμαστε μια έκθεση η οποία να χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο κοινό μα στόχο. Σε σχέση με τι δύο τελευταίε παρεμβάσει που έγιναν, δεν ξέρω ε, κατά πόσο μπορώ να συμφωνήσω. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό που είπε η Περβάνς. Ε, γίνεται ένας τεράστιος αγώνας ε, εκ μέρου των παραγόντων της δημοσιονομικής πολιτικής, οι οποίοι λένε ότι η άμυνά μας είναι να πούμε ότι όσον αφορά το δημόσιο χρέος δεν υπήρχε αρκετή δημοσιονομική πειθαρχία. Εγώ θεωρώ ότι το δημόσιο χρέος βεβαίως ε, θα πρέπει να συνοδεύεται από τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις. Αλλά θα φτάσουμε σε μια εξυγίανση μόνο εφόσον εμπλέξουμε και τους εργαζόμενους σε αυτή τη διαδικασία. Και έχει δίκιο η τα λέει ότι υπάρχουν αγώνες που δεν ε, παίζονται σε ε, χώρες άλλες όπως είναι η Ιαπωνία. Ενώ σε εμά γίνεται μια συνεχής προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ευρωζώνης. Ακόμα και σε χώρες που έχουν υψηλό χρέος. Δεν, γίνεται, δεν γίνονται ίδιες επιθέσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ερμηνεύσουμε σωστά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως είπε η γιατί έχουν γίνει πολλές ερμηνείες, αλλά δεν ε, τηρούνται τα κριτήρια. Και η Γαλλία και η Γερμανία παραβίασαν αυτά τα κριτήρια. Και είπαν ότι και εμείς έχουμε δημόσια χρέη, αλλά δεν θέλουμε καμία επιβολή κυρώσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε ότι να υπάρχουν ξεκάθαρες δομές. Η Περβάνς γράφει ότι το σύμφωνο σταθερότητα έχει έναν κατασταλτικό, καταπιεστικό χαρακτήρα. Και στη γαλλική μετάφραση αναφέρεται αυτό ρητά. Αν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, ούτω ώστε να εφαρμοστούν τα μέτρα και να πούμε ότι θα πρέπει να τηρήσετε τα συμφωνηθέντα κριτήρια, θα πρέπει να μεριμνήσετε για μια λελογισμένη χρήση των κονδυλίων, μόνο τότε έχουμε μια σωστή πιθανότητα. Δεν είμαι υπέρ του να τροποποιήσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, αλλά θεωρώ ότι το Σύμφωνο Σταθερότητα έχει μία ευκαιρία μόνο εφόσον συνοδεύεται από μία σωστή παρακολούθηση και μία εφαρμογή μηχανισμών που ε, ακριβώς ελέγχει την πειθαρχία στο επίπεδο των εργοδοτών και των εργαζομένων. Ευχαριστούμε πολύ. Στην έκθεση ε, γίνονται κάποιες προτάσεις που έχουν μια επίπτωση στην Κομισιόν. Γι' αυτό η Κομισιόν παρακάλεσε να πάρει και αυτή το λόγο. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σφίμπαντ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση ε, Ανταγωνιστικότητα. Είμαι υπεύθυνη για τα θέματα αυτή, αυτά μεταξύ άλλων, καθώς επίσης και για την απάτη για τις ε, ε, οικονομικές υπηρεσίες. Εγώ κυρίως θα σας μιλήσω για τα θέματα του ανταγωνισμού, αλλά είμαι βέβαιη ότι οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Market ε, θα έχουν πράγματα να σας πούνε και μπορούμε να σας δώσουμε και σχόλια γραπτός. Αυτό που θα ήθελα να κάνω εντάχει είναι να σας πω καταρχάς ότι λυπάμαι ότι, γιατί προσφερθήκαμε επανειλημμένως να έρθουμε να εξηγήσουμε το ρόλο της πολιτικής ανταγωνιστικότητας και οι δράσεις που λάβαμε και λαμβάνουμε ακόμα στον τομέα της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν έχουν ληφθεί υπόψη. σχόλιο εκτό μικροφώνου. Το ξέρω, αλλά ορισμένε φορέ σε τεχνικό επίπεδο ίσω θα έπρεπε να προσπαθήσετε να κατανοήσετε λίγο τι ε, δυσκολίε, ε, διότι διαβάζοντα την έκθεση, κάποιε διευκρινήσει που θα σα είχαμε δώσει μπορεί να ήταν χρήσιμε για σας. Θα μπορούσα κάλλιστα βέβαια να σας δώσω και τα σχόλια αυτά γραπτός, με μεγάλη μου χαρά μάλιστα. Ένα από τα σχόλια που θα σας αποστείλουμε γραπτός είναι το 149, ο έλεγχος των συγχωνεύσεων, γράφεστε ότι δεν ε, υπάρχει τομέας τη πολιτική ανταγωνισμού για να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, οργάνωση των back office, επενδυτικές τράπεζες ε, και ούτω καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το, την εξουσία για να ε, δει τι γίνεται με τις συγχωνεύσεις σε όλους τους τομείς και στις επενδυτικές τράπεζες και στην οργάνωση του back office και των δραστηριοτήτων, ε, των ε, οίκων αξιολόγηση κλπ. Όλα αυτά θεωρούνται συγχωνεύσεις βάσει του κανονισμού για τις συγχωνεύσεις και έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, ακόμα και αν ο κίνδυνος προκύψει ε, στον τραπεζικό τομέα. Αυτά ελέγχονται στο σχετικό κανονισμό και τα μέλη, τα συμβαλόμενα στη συγχώνευση δεν μπορούν προχωρήσουν χωρίς έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν δημιουργηθεί ή ενισχυθεί μια κυρίαρχη θέση, δεν επιτρέπονται οι, οι μπορούν να απαγορευτούν ή αν θεωρηθεί ότι υπάρχει στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Το έχουμε κάνει αυτό. Για παράδειγμα, η αγορά της BNP Paribas ή της ε, φορτή ε, του Βελγίου και τη φορτή του Λουξεμβούργου ελέγχθηκε βάσει του κανονισμού των συγχωνεύσεων. Ε, Έχουμε δει τι γίνεται με την BNP ε, Paribas ε, για, το, ε, για την καταναλωτική πίστη στο Βέλγιο και ελέγχεται και το θέμα των πιστοτικών καρτών και του Λουξε, της τράπεζας του Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Έχουν ληφθεί μέτρα λοιπόν και να πω ότι και στον έλεγχο των κρατικών επιδοτήσεων και στα διαρθρωτικά ταμεία κάθε φορά που ζητούνται επενδύσεις πάντα φροντίζουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι επενδύσεις δεν θα μας οδηγήσουν σε μια κατάσταση που θα είναι κατά της ανταγωνιστικής ε, αλλά σε μια κατάσταση που θα είναι υπέρ τη αγωνιστικότητα. Αυτό είναι και ο λόγο ύπαρξή μα εδώ. Ε, μπορεί να υπάρχουν κατόφλια που δεν μας επιτρέπουν να παρέμβουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές επαφέ με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να δείξω είναι αυτό που έχετε στο σημείο 88. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία πρόταση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή της κρίσεως υιοθέτησε πότε να σας πω τώρα, στο πρώτο τμήμα, στο πρώτο εξάμεινο, ένα πακέτο μέτρων τα οποία προκύπτουν από ανακοινώσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτέ οι ανακοινώσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και δίνουν και κατευθυντήριε γραμμέ προ τα κράτη-μέλη όσον αφορά την αξιολόγηση και την ανταγωνιστικότητα των μέτρων υποστήριξης για τις ε, τράπεζες και την πραγματική οικονομία. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, μοντέλα αποζημιώσεων για τον τραπεζικό τομέα και υπάρχουν και μέτρα για την πραγματική οικονομία. Τα μέτρα για το χρηματοπιστωτικό τομέα διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα υποστήριξη τα οποία δίνονται από τα κράτη-μέλη, παρά το γεγονό ότι δεν είναι αρμονισμένα, αυτό το δεχόμαστε, αλλά δεν έχουν όλοι το ίδιο σύστημα στα κράτη-μέλη, μας έδωσαν όμως τη δυνατότητα να έχουμε ένα μέσο συντονισμού για τα εθνικά συστήματα υποστήριξης, κυρίως ως προς την τιμολόγηση των εγγύσεων και κίνητρα για να ε, επιστραφεί το κρατικό κεφάλαιο, ρήτρε ε, ω προ τι αποζημιώσει και ένα από τα βασικά στοιχεία αυτών των εθνικών προγραμμάτων ήταν να διασφαλίσουμε ότι μπορούν οι τράπεζε να συνεχίσουν να δανειοδοτούν την πραγματική οικονομία. Γι' αυτό ακριβώ και αλλάξαμε την προσέγγιση μα στην ανακοίνωση για την ε, επανακεφαλαίωση, για να μπορέσουμε ε, να δούμε τι γίνεται με τι πιο υγιεί και τι λιγότερο υγιεί τράπεζε. Επομένω, να μην υπάρχουν οι ίδιε προποθέσει για τι υγιεί και μη υγιεί τράπεζε. Νομίζω ότι όλα αυτά λοιπόν ήταν μέρος μιας διαδικασίας όπου υπάρχει συνεχής συντονισμός και διασφαλίζουμε ότι τα εθνικά συστήματα υποστήριξης έγιναν με συντονισμένο τρόπο. Και υπάρχουν και μηχανισμοί συντονισμού και για τις κρατικές ε, επιδοτήσεις, να μην υπάρχουν φαινόμενα στρέβλωσης του ανταγωνισμού και ε, οι τράπεζες να αναλάβουν και τμήμα της ε, διάσωσής τους. Υπάρχουν κάποιοι επιπλέον περιορισμοί όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Ακριβώς και για να είναι καταμερισμένο το κόστος ε, των κονδυλίων τα οποία πρέπει να επιστραφούν ε, Υπάρχουν μέτρα για τις πληρωμές, έχουν συμπεριληφθεί και στα προγράμματα αναρθοδιάθρωσης τα οποία έχουμε δεχτεί και την αναθεώρηση του συστήματος αποζημίωσης, ε, θέματα ε, επιχειρηματικής διακυβέρνησης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία εξετάζουμε όταν ε, ε, γίνεται έλεγχος για τις κρατικές επιδοτήσεις. Τώρα, στο σημείο που μιλάτε για την έξοδο. Νομίζω ότι από την αρχή της κρίσης είχαμε πάρα πολλές τράπεζες ε, το φαινόπωρο του 2008 που ζητούσαν να τη σώσουμε και ε, ήταν σαφές ότι δεν θέλαμε να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπως στις ΗΠΑ με τη Lehman Brothers και να μην έχουμε μεγάλη κατάρρευση επιχειρήσεων και φυσικά όλο τον κίνδυνο ο οποίος προερχόταν ε, από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ίσως είμαστε πάρα πολύ ελαστική για τη διάθεση των τραπεζών, αλλά από την αρχή είπαμε ότι θα φτάσει μια στιγμή που θα πρέπει να πληρωθεί ένα αντίτιμο για όλα αυτά και η αναδιάθεση των τραπεζιών που έλαβαν κρατική επιδότηση θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες και αυτό φυσικά για τις επιχειρήσεις με τις οποίες έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας σημαίνει ότι είχαν πάρα πολύ σημαντική μείωση του ισοζυγίου τους διότι ακριβώς λήφθη αυτό το στοιχείο υπόψη. Ήταν σαφές λοιπόν από την αρχή ότι θα φτάσει κάποια χρονική στιγμή στην οποία τα εξαιρετικά μεγάλα ποσά τα οποία δόθηκαν στον τραπεζικό τομέα θα επιστραφούν. Ε, τονίζαμε πάντα από την αρχή ότι οι κανόνες που εφαρμόζουμε είναι εξαιρετικοί κανόνες, είναι μια ειδική εξαιρετική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έχουμε μια συγκεκριμένη νομική βάση, μια νομική βάση που... Ε, ξεκινά από τη σοβαρή στρέβλωση στις αγορές των κρατών μελών και για να επανέλθουμε στην ομαλότητα θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα, αλλά χρειαζόμαστε μια νέα κατάσταση ομαλότητα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη και την κατάλληλη διακυβέρνηση και την κατάλληλη διαχείριση. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι εν αυτή τη στιγμή ε, στι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα σα κάνουν οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Μάρκετ. Τώρα, η διαδικασία του phasing out, η επιστροφή στην ομαλότητα, ήταν κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί από την αρχή. Ο κύριο Αλμούνια φαντάζομαι ότι το είχε ε, επισημάνει. Είμαι βέβαιη ότι το είχε επισημάνει, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ακόμα υπάρχουν κίνδυνοι στι χρηματοπιστωτικές αγορέ, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε στα φυσιολογικά πλαίσια. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που ε, ξεκινήσαμε ήταν το phasing out των προγραμμάτων εγγύησεων. Δηλαδή, από 1η Ιουλίου του 2010 και μετά θα αρχίσουν να είναι πιο υψηλές οι τιμές, ε, θα σχετίζονται περισσότερο με την ε, πιστοτική αξιοπιστία των τραπεζών που συμμετέχουν σε αυτά τα συστήματα εγγυήσεων, που σημαίνει ότι ενθαρρύνουμε τις τράπεζες που είναι ακόμα μέσα στο σύστημα να φύγουν από το σύστημα και επίσης τις τράπεζες που δεν έχουν τρόπο ε, ακόμα να φύγουν, να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα και επομένως σημαίνει ότι σας λέει η Κομισιόν ότι αν δεν είστε έτοιμοι να βγείτε πρέπει να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες και το ίδιο θα κάνουμε και για τα προγράμματα ε, για τα κεφάλαια. Πρέπει να δούμε τις ίδιες συνθήκες. Εδώ βέβαια τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, διότι σε αυτά τα προγράμματα ήδη έχουμε ενσωματωμένες προϋποθέσεις με διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σταδιακά και επομένως προς το παρόν εστιάζουμε στα προγράμματα εγγύησεων. Τέλος, στην παράγραφο 149 ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει τι θα γίνει με τις επενδυτικές τράπεζες. Ε, αυτό δεν είναι κάτι καινοφανές. Ε, το έχουμε εξετάσει και το εξετάζουμε και εξετάζουμε τις τράπεζες επενδύσεων για να δούμε αν υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με τους κανόνες ανταγωνιστικότητας του άρθρου 101 και άρθρου 102 που σημαίνει ότι έχουμε ε, παράνομες συμφωνίες ή ε, μη ανταγωνιστικές θέσεις. Ναι, μεν ε, μιλούν από θέση ισχύω, αλλά είναι πολύ περιορισμένη αυτή η θέση. Ε, μπορεί να ανοίξει μια τέτοια υπόθεση αν όντω υπάρχουν ενδείξεις ε, ότι κάποιος συγκεκριμένο συγκεκριμένος ο οποίος συμμετέχει στην αγορά δεν συμμορφούνται προς τους κανόνες ανταγωνιστικότητας. πρέπει να το εξετάσουμε, δεν λέω ότι δεν το εξετάζουμε, αλλά δεν έχουμε κανόνες που μας επιτρέπουν απλώς να επιτεθούμε σε κάποιον, ε, σε δομές ε, οι οποίες είναι κατά της ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφή συμπεριφορά που είναι κατάχρηση της προεξάρχουσας θέσης. Η προεξάρχουσα θέση αυτή καθεαυτή δεν αποτελεί τεκμήριο για κάτι τέτοιο. Εξετάζουμε ακόμα τον τομέα αυτό όχι μόνο τις επενδυτικές τράπεζες αλλά και τους οίκους αξιολόγησης και όλους τους υπολείπους ε, όλο αυτό το τοπίο το οποίο αφορά όλο το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Δεν λέω ότι αποφεύγουμε τις ευθύνες μας και μιλησουμε Ίσα ίσα είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να αναλάβουμε μέτρα, αλλά ε, υπάρχουν περιορισμοί στους κανόνες μας και το Δικαστήριο και το Ευρωκοινοβούλιο είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα μας βάλουν τις φωνές άμα ξεπεράσουμε τα όρια μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσαμε να λάβουμε κάτι γραπτό από εσά και από του ε, συναδέλφου σα. Ε, θα σα παρακαλούσα να λάβετε υπόψη στο το χρονοδιάγραμμά μα, ε, ώστε να έχουμε το χρόνο να εξετάσουμε τα έγγραφά σα εγκαίρω. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι στο Κοινοβούλιο αρκετό καιρό και είναι σαν ένα μεγάλο χωνευτήρι και όλα όσα βγαίνουν είναι γκρίζα, διότι πρέπει να επιτευχθεί συνένεση για όλα τα θέματα. Και ένα από τα πλεονεκτήματα της πολιτικής είναι ακριβώς ότι ε, υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Ε, γι' αυτό έγινα μέλος του πολιτικού μου κόμματος πριν πάρα πολλά χρόνια. Ε, είναι πάντα χρήσιμο να καταλήγουμε σε συνένεση, αλλά είναι και χρήσιμο να βλέπουμε πού υπάρχουν οι διαφορές των απόψεων. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι συναρπαστικό το έγγραφο αυτό. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Θυμάμαι τότε που ήμουν εγώ πάντα στην αντιπολίτευση ε, και ε, ε, έκανα αντιφάσεις, αλλά δεν θα το κάνω αυτό σήμερα. Πιστεύω ότι όπως και στα παραμύθια θα καταλήξουμε σε, σε μια συνένεση, αλλά το ότι η κυρία Περές εκπώνησε την έκθεσή της δίνει στους υπολείπους από εμάς, τουλάχιστον δίνει σε μένα τη δυνατότητα να Ε, ξανασκεφτώ λίγο τις θέσεις μου και να επανέλθω στις θέσεις των σοσιαλδημοκρατών ε, που πάντα κυριαρχούσαν στη χώρα μου. Νομίζω ότι καταρχήν θα πρέπει να πούμε τι θα αποκομίσει το κοινό από την έκθεση αυτή. Θα μπορούσαμε να πούμε σε λεπτομέρειες όπως κάνανε κάποιοι από εσά. Ε, μπορούμε να κάνουμε πολλές τροποποιήσεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες. Πριν πολλά χρόνια όμως ε, ήμουνα ε, ανταποκριτής δημοσιογράφος και διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διάβαζαν αυτά που έγραφα, διάβαζαν τον τίτλο και γι' αυτό θα πρέπει όλα να συμπεριλαμβάνονται στον τίτλο. Ο τίτλος μου και ελπίζω η πολιτική μου ομάδα να με ε, υποστηρίξει αλλά με του φιλελεύθερου ποτέ δεν ξέρει κανείς. Εμένα ο τίτλος μου θα ήταν ε, «Το παγκόσμιο μοντέλο της ελεύθερης αγοράς ε, και του ελεύθερου εμπορίου επιβίωσε την χειρότερη κρίση από το 1930». Και ακριβώς αυτό είναι το σημείο κίνησής μου, αυτή είναι η βάση μου. Φυσικά πρέπει να ομολογήσουμε ότι, έχουμε γίνει, ότι έχουν γίνει πολλά λάθη. Και πρέπει να ασχοληθούμε με τα λάθη αυτά και ακριβώ αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τελικά όμως, η κρίση αυτή δείχνει ότι η μόνη εναλλακτική λύση για να έχουμε ευημερία και αξιοπρεπή ζωή όσο γίνεται περισσότερου ανθρώπου στον κόσμο, είναι το μοντέλο που έχουμε. Μπορεί να το ονομάσει κανεί ε, το μοντέλο τη κοινωνική αγορά. Ε, εγώ, ε, ω φιλελεύθερο, ε, λέω ότι είναι ένα κοινωνικοφιλελεύθερο μοντέλο ευημερία. Ε, έχουμε φυσικά κάποιες διαφωνίες μεταξύ μας αλλά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε τελικά σε συνένεση. Η ομάδα μας ε, πιστεύει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και θα συμφωνούσαμε αυτό. Δεν ε, έπιασα όλες τις παραγράφους που αναφέρατε, αλλά με πολλές από αυτές δεν έχουμε πρόβλημα. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Όσο περισσότερη Ευρώπη προτείνουμε όμως, τόσο περισσότερη νομιμότητα χρειαζόμαστε από την κοινή γνώμη. Και θα σας στηρίξουμε στο ζήτημα αυτό. Σχετικά με τα όσα έχουν γίνει, κύριε Περέζ, δεν θα σας εκπλήξει ότι έχουμε να προτείνουμε κάποιες διαφορετικές διατυπώσεις, ε, θα επιλέγαμε και διαφορετική δομή στο κείμενο. Εξετάζοντας όμως το τι έχει γίνει και αυτό που συζητάνε όλοι αυτή τη στιγμή, την περίπτωση της Ελλάδας δηλαδή, πιστεύω ότι οι χώρες του Νότου μπορούν να ακολουθήσουν αυστηρούς κανόνες όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε σε μια απόλυτα ειλικρινή έρευνα τι πήγε στραβά. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε από εδώ από τράγους. Θα βρούμε τόσο πολλούς που δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Το κοινό απαιτεί όμως να βρούμε τι πήγε στραβά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήξερε τίποτα, άλλα θεσμικά όργανα, η Κομισιόν, κάποια μέλη του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Δεν θα πρέπει όμως ε, να καταλήξουμε σε, ε, ε, σε δημαγωγικές πρακτικές, να αναφέρουμε ονόματα και να τους κατηγορούμε. Ναι, εδώ είμαι, <laughs> λέει ο μιλητής. Κυρίως ήταν πολιτικά τα λάθη που έγιναν. Θα πρέπει να είμαστε ακριβείς ως προς τα θέματα αυτά και μία από τις συστάσεις της έκθεσης θα πρέπει να είναι να συσταθεί μια πολύ αυστηρή ομάδα έρευνας. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το κάνει αυτό και δεν θα πρέπει να ντραπούμε αυτά που πιστεύουμε, να πούμε τι πήγε στραβά και να προτείνουμε κάποιες αλλαγές. Κυρία Περές, λοιπόν, είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ε, ελπίζουμε πάντως ε, η πλειοψηφία να στηρίξει τη θέση των φιλελευθέρων. Θέλουμε να πετύχουμε μια ευρεία συνένεση Με βάση αυτά που γράψατε στην έκθεσή σας, ελπίζω ότι θα ακούσετε τη θέση μας ε, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να ε, ξεφύγουμε από την κρίση αυτή. Διότι το μήνυμά μας, αυτό που θα λέμε τελικά, τα συμπεράσματά μας, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον τίτλο, στην αρχή της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από κάποια θέματα ε, φόρμα, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γιατί νομίζω ότι η μέθοδο είναι ιδιαίτερω καθοριστική για μια ποιοτική εργασία. Την τελευταία φορά στο Στρασβούργο, όταν παρουσίασε Περβάν στην έκθεσή τη, είπαμε όλοι ότι όσον αφορά τη φόρμα θα πρέπει να βρούμε μια λύση ούτως ώστε η έκθεση να είναι πιο εύληπτη, πιο ευανάγνωστη. Και τέθηκαν ορισμένες ε, ερωτήσεις δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να δοθούν κάποιες απαντήσεις σήμερα, ε, γιατί αν ε, είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε αυτή τη φόρμα που επιβάλλει το Κοινοβούλιο, να μπορέσουμε να έχουμε ένα κείμενο το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει που ανέφερε ο Όλε Σμιτ όσον αφορά την, ε, το ευανάγνωστο, την ευληπτότητα, δηλαδή τους πηχαίους τίτλους. θέσαμε λοιπόν το ερώτημα αυτό. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα και να έχουμε μία απάντηση. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο αφορά τους, ε, την ενημέρωση των αριθμών ε, και των συμβάντων, γιατί διδραματίστηκαν πολλά τις τελευταίες εβδομάδες και μου φαίνεται λογικό όσον αφορά την ποιότητα ένταξης αυτών των νέων στοιχείων στην έκθεση ε, να το κάνει, να το πράξει υπερβάνω, να συμπεριλάβει δηλαδή αυτά τα καινούργια στοιχεία. Αλλά Εάν το κάνει υπό το πνεύμα του δικού της οράματος, νομίζω ότι θα δείχνουμε σε συγκρούσεις. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι η συγγήτρια θα μπορούσε να κάνει αυτή την εργασία αντικειμενικής συμπερίληψης όλων των ε, στοιχείων. Ε, και θα ήθελα να μου δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση επί τούτου, κατά πόσο προτίθεται να το κάνει. Τώρα, Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ε, θέτει εμφαντικά η έκθεση ως επιθυμίες. Μιλάει για τις διάφορες ε, αναλύσεις, διαφορετικές αναλύσεις ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχουμε θέσει εδώ και πολλούς μήνες. Στην ε, ανακοίνωση της ΡΕΝ πριν από μερικά μερικές εβδομάδες γίνεται σχετική αναφορά. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτό το σημείο. Γιατί το κείμενο αυτό, η έκθεση αυτή εγγράφεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ορισμένες φορές οι προτάσεις μας την χάνουν της συμφωνίας και του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Τώρα, το τελευταίο σημείο της παρέμβασής μου αναφέρεται σε αυτό το οποίο είπε ο Όλε Σμιτ με με τι θέλουμε να έχουμε στο τέλος. Υπάρχουν δύο σκόπελοι που θα πρέπει να αποφύγουμε. Ο πρώτος είναι ένα διπλωματικό κείμενο που λέει τα πάντα και το αντίθετό τους. Το δεύτερο, ο δεύτερος σκόπελος είναι ένα κείμενο ε, συσχετισμού δυνάμεων όπου υπάρχουν διάφορα μπλοκ ε, και τελικά γίνεται η ψηφοφορία. Όπως έγινε για παράδειγμα στην έκθεση Βαντόκ. Ε, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, μπορεί να γίνουν τα πάντα, δηλαδή στη βάση του σχετισμού δυνάμενα να γίνει ψηφοφορία. Εγώ είχα προτείνει τότε, αλλά δυστυχώς δεν με άκουσαν εδώ και πολύ καιρό, να μπορούμε να επικεντρωθούμε γιατί είναι μεν οι συζητήσει αυτέ είναι ενδιαφέρουσε, αλλά αν ο καθένα παρουσιάζει το δικό του πρόγραμμα και κάποιος λέει θέλω πιο πράσινη πολιτική, περισσότερο περιβάλλον κλπ. Ο άλλος λέει πιο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Δεν είναι αυτό το οποίο θα στηρίξει την ποιότητα του τελικού συμβιβασμού. Νομίζω σημαντικό είναι να, ίσως να σχηματιστούν πιο μικρές επιτροπές ή να συνέλθουν μικρότερες επιτροπές και να ε, εντοπιστούν σχέση σημεία κλειδί επί των οποίων θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε συνένεση. Για παράδειγμα, η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμιοποίησης. Ο καθένας μπορεί να υποβάλει τις δικές του τροπολογίες, ο Όλε Σμιτ θα υποβάλει μια τροπολογία για το διεθνές εμπόριο ως ε, ίστατο στόχο και λοιπά, ως μέσο ειρήνευση των λαών. Άλλοι θα έχουν προστατευτικούς στόχους, άλλοι ρυθμιστικούς κλπ. Και δεν θα κατορθώσουμε να οικοδομήσουμε εδώ κάτι το οποίο ε, αποτελεί στοιχείο αναπόσπαστο της κοινή ε, της δημόσιας συζήτησης και το οποίο περιμένουν οι πολίτες. Κανείς δεν θέλει να πάει προς μια προστατευτική κατεύθυνση από τη μία, από την άλλη. Δεν είναι δυνατόν από μόνοι μας να κάνουμε ελεύθερες συναλλαγές αν οι υπόλοιποι δεν το επιθυμούν. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται κατ' επανάληψη στα κείμενα επί των οποίων ε, εργαζόμαστε, στην ΕΚΟΝ για παράδειγμα, για τα, για τα Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων. Αυτό το ζήτημα είναι στην καρδιά του προβλήματος και προσπαθούμε να, βρούμε μια πλειοψηφική λύση που συμμερίζεται αυτή τη στιγμή ένα τμήμα των φιλελευθέρων, γιατί είναι δύσκολο να κερδίσει κανείς το σύνολο των φιλελευθέρων. Εγώ θα ήθελα να πάρουμε σαν βάση αυτή τη θέση και αν είναι δυνατόν να υπάρξει ένας εφικτός συμβασμός, ίδιες υποχρεώσεις, ίδια καθήκοντα. Δηλαδή, ανοίγουμε την ευρωπαϊκή αγορά σε παράγοντες που βρίσκονται παντού στον κόσμο, μπορούν, αλλά δεν μπορούν να εμπορευθούν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά παρά μόνο εφόσον τηρούν κάποιους κανόνες που είναι αυτοί που εφαρμόζονται για τους Ευρωπαίους. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βρούμε διάφορες αποχρώσεις ε, διαφορετικές. Αλλά νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να τοποθετηθεί όχι μέσω της μάχης των τροπολογιών που τελικά δεν μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε έναν συμβεβασμό. Τώρα, τα όσα είπε ο κύριος Μαν όσον αφορά τη συζήτηση εν σχέση ε, με την, ε, το σεβασμό, την τήρηση του συμφώνου σταθερότητα από τη μία και ανάπτυξη από την άλλη. Δηλαδή τη σύντηση μεταξύ λιτότητα, μέτρο λιτότητα και οικονομική ανάπτυξη από την άλλη. Έτσι τίθεται στην Γαλλία μα στου όρου. Και από τη στιγμή που ένα τμήμα των κινδύνων που συνδέονται με το δημόσιο χρέο είναι ε, θεωρούνται ε, ασφαλίζονται, θα πρέπει το ίδιο να γίνει και με τον έλεγχο. Γιατί εάν μειωθεί το δημόσιο χρέος ενός ε, κράτους, ε, λέχθηκε ότι θα πρέπει οι επενδύσεις να ανακάμψουν, αλλά οι επενδύσεις δεν είναι δυνατόν να ανακάμψουν ε, σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρχίσουν οι επιχειρήσεις να επενδύουν μαζικά. Είναι παράλογο από οικονομική άποψη. Ε, είμαστε εμείς σε θέση να το κάνουμε γιατί οι χώρες πρέπει να βρουν κάποιους συμβασμούς. Είμαστε σε θέση εμείς με τις διαφορετικές μας προσεγγίσεις, με διαφορετικέ διαφορετικές προτεραιότητες είμαστε σε θέση να εξάγουμε αυτό το συμβασμό ή θα πρέπει να αρκεστούμε, όπω είπα, σε μία μάχη των τροπολογιών και σε σχηματισμού δυνάμεων. Εμένα θα μου άρεσε η Επιτροπή αυτή να εξυπηρετήσει ακριβώς αυτό το στόχο. Δεν έχω την εντύπωση ότι κινούμεθα σε αυτό το δρόμο. Ο Σταύρος κ. Καράς είπε «εντάξει, να πάρουμε άλλη μια εβδομάδα, αλλά υπό την προπόθεση να γίνει μια ποιοτική εργασία εντός αυτής της εβδομάδας, όχι μόνο ακόμη μια εβδομάδα για να κάνουμε τη μάχη, να δώσουμε τη μάχη των τροπολογιών. Νομίζω ότι οι συνοριστές θα πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτή τη γραμμή και να προσπαθούν να βρουν έξυπνες συμβαστικές ε, λύσεις. Thank you very much, Mr. And... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την Περβάντς ε, για όλη τη δουλειά που έχει κάνει για το θέμα αυτό. Από πού να αρχίσω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο με ένα έγγραφο στο οποίο κάποιος έχει δώσει την ψυχή του να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ ε, των προσωπικών μας πεπιθήσεων και της ερμηνείας των γεγονότων. Ε, φαντάζομαι ότι αν το είχα γράψει εγώ θα ήταν τελείως διαφορετικό κείμενο το οποίο θα προέκυπτε ακριβώς από τα ίδια στοιχεία και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για όλους τους παρισταμένους εδώ στην αίθουσα. Αντί να διατρέξουμε την έκθεση και τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν, νομίζω ότι θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Πασχάλ. Πώς θα προχωρήσουμε. Διότι δεν νομίζω ότι Αρκεί το γεγονό ότι ο καθένας από εμά θα ξαναέγραφε την ίδια έκθεση με τα ίδια γεγονότα και με τα ίδια συμπεράσματα. Καλό θα ήταν ίσω να βγάλουμε λίγο τις πολιτικές από μέσα, διότι υπάρχουν κάποια συμπεράσματα με τα οποία ίσως δεν θα συμφωνούσαν πολλοί από εμά εδώ στην αίθουσα, αλλά να δούμε ποια είναι τα κύρια αίτια, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των αιτίων και ε, από εκεί και πέρα σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι σαφές ότι στην έκθεση αυτή έπρεπε να δούμε ποια είναι τα πραγματικά αίτια και ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα της πολιτικής που θα προκύψουν από αυτά. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Όταν το δίνω σε κάποιον να το διαβάσει, πραγματικά δεν ξέρουν σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε. Επομένως, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν άλλο μηχανισμό, όπως όλοι είπανε, για να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη εκδοχή που θα δοθεί στο κοινό. Ε, φαντάζομαι να ε, καταλήξουμε σε αυτή πριν κάνουμε τις συμβαστικές συζητήσεις. Πραγματικά δεν ξέρω τι μέρο γενέστε με αυτό το πράγμα. Ε, υπάρχουν πολλοί εδώ, πολύ πιο εμπειροί από μένα που μπορούν να μας πούνε τι ακριβώς θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά το να ξανακαθίσουμε και να γράψουμε άλλη έκθεση σίγουρα δεν θα μας βοηθήσει γιατί θα έχουμε άλλες ε, χίλιες τόσες τροπολογίες και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση θα εκραχυνθεί. Ε, καλό θα ήταν από σήμερα κιόλα να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες σε αυτή την έκθεση, είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό και το να προσπαθήσουμε να το τροποποιήσουμε πραγματικά θα ήταν ε, κρίμα διότι θέλουμε μια έκθεση την οποία ναι μεν να δεχόμαστε όλοι από πολιτικής πλευράς αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τη χάραξη της πολιτικής μας από εκεί και πέρα. Ε, στο παρελθόν δεν υπήρχε κανένας πιο επικριτικός από μένα για τις επενδυτικές τράπεζες. Αλλά το να λέμε ότι αυτές φταίνε χωρίς να έχουμε κανένα στοιχείο ε, που να το αποδεικνύει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες και υποθέσεις ανά τον κόσμο, αλλά πολύ λίγες υποθέσεις έχουν καταλήξει στο δικαστήριο. Όταν κάνουμε λοιπόν τέτοιους ισχυρισμούς, καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ε, με λυπεί κάτι που διάβασα εδώ στην έκθεση, στο σημείο 181. Έλαβα τόσα πολλά τηλεφωνήματα για τη συγκεκριμένη αυτή φράση από δημοσιογράφους και πραγματικά δεν είναι και μόνοι αυτοί οι οποίοι μου τηλεφώνησαν, είναι και πάρα πολλοί φίλοι που μου τηλεφώνησαν και μου λένε το ίδιο πράγμα. Πώς θα καταλήξουμε λοιπόν σε ένα τελικό έγγραφο, πραγματικά δεν ξέρω. Στο 206 που μιλάμε για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Η κινητικότητα είναι κάτι για τους πολύ πλούσιους και για τους πολύ πτωχούς. Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί στην περιφέρειά μου θα σας πούμε ότι δεν ισχύει. Έχουμε τεράστια κινητικότητα από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα λοιπόν να πιστέψω αυτή τη δήλωση όταν στην ίδια μου τη χώρα το 60% των αιτήσεων ε, για ε, φίτηση στα πανεπιστήμια μας είναι από ε, άλλες χώρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουν και να σχετιστώ με αυτή τη δήλωση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να φύγει από το κείμενο η πολιτική έμφαση και να μείνουμε στα συμπεράσματα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι ε, πολύ απτό. Βέβαια είμαι βέβαιη ότι η υπερβάνηση θα μας βοηθήσει να βρούμε τη λύση. to be... Μου φαίνεται ότι έχουμε έναν γύρο επικοδομητικών σχολείων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι άσχετα από το τι μπορεί να πιστεύει ο κόσμος όταν συζητάει την έκθεση στην ομάδα του, θέλουμε να καταλήξουμε σε μία ισχυρή έκθεση με ισχυρά μηνύματα. Υπάρχει ήδη ουσία στα μηνύματα κλειδιά της έκθεσης αυτής. Επειδή η έκθεση προσπαθεί να συμπεριλάβει την ανάγκη για νέες επενδύσεις, για ρύθμιση, καθώς και ανακατανομή ε, της οικονομίας και πιο πράσινη οικονομία, υπάρχει πολύ ουσία στα βασικά μηνύματά της. Υπάρχει λοιπόν βάση για συνένεση που να ξεπερνά τα όρια των πολιτικών ομάδων εδώ στην, στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο. Δεν θα επαναλάβω τα σημεία όπου συμφωνούμε με την εισηγήτρια. Θα αναφέρω τα σημεία όπου έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Ένα από αυτά είναι το σημείο κλειδί για οποιονδήποτε πράσινο το πώς η περιβαλλοντική κρίση εντάσσεται στο όλο πλαίσιο. Η περιβαλλοντική κρίση είναι κυρίως κοινωνική, αν την εξετάσει κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλο και περισσότεροι θέλουν παρόμοιο βιωτικό επίπεδο με μας. Και γι' αυτό εξαντλούμε τους πόρους. Είναι λοιπόν πολύ περισσότερο κλιματική είναι κάτι πολύ περισσότερο από κλιματική κρίση. Είναι κρίση που έχει να κάνει με τη χρήση της γης, με τους πόρους, με την τιμή τους και γι' αυτό είναι η οικονομική κρίση και συνδέεται και με την κρίση της βιοποικιλότητας. Γι' αυτό η περιβαλλοντική κρίση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προοπτική βορρά-νότου η προοπτική αυτή είναι πολύ λιγότερο γεωγραφική σήμερα. Είναι θέμα ενέργειας και κλίματος, είναι όμως γενικά θέμα υπερεκμετάλλευσης του πλανήτη σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό, όσον αφορά την πράσινη οικονομία, θα πρέπει να εξετάσουμε θέματα πέρα από την ενέργεια, την αποτελεσματικότητα των πόρων, το κεφάλαιο υλικού πλούτου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι και θέμα τεχνολογίας. Πόσος είναι ο όγκος του κεφαλαίου αυτού και πόσο, πόση χρήση είναι δυνατόν να γίνει από αυτό το κεφάλαιο. Για να προχωρήσουμε λοιπόν σε μια πιο ισχυρή προοπτική στην εκθεσία αυτή θα πρέπει να εξετάσουμε τι σημαίνει η πράσινη οικονομία για τους τομείς που θα πρέπει να οδηγήσουν σε ανάπτυξη των, σε αύξηση των θέσεων εργασίας στο μέλλον. Χρειάζεται να γίνει μια μετατροπή της οικονομίας και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα ήταν καλό να εμπλουτιστεί με κάποιες τροπολογίες που να συμπεριλαμβάνουν ε, την πτυχή των δύο φύλων στην κρίση. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τις αιτίε της κρίσης, υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε. Στα σημεία 32 και 33, που είναι σημεία κλειδιά. όσον αφορά την κατανόηση του τι προκάλεσε την κρίση. Πιστεύω από τη μία ότι είχαμε μια απότομη αύξηση του φθηνού χρήματος. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα της, διά, της διάκρισης στην εξήγηση, ότι στη φούσκα αυτή του χρήματος ε, μέρος των χρημάτων ήταν καλό και μέρος ήταν κακό. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον εάν εξετάζαμε ε, σε, στο ίδιο επίπεδο τις διάφορες ε, πηγές της κρίσης. Υπάρχουν κάποιες ανισότητες και ανισορροπίες που οδήγησαν σε αυτή τη φούσκα χρήματος. Από την άλλη, η λεγόμενη πολιτική αριστερά θα πρέπει να, εξετάσει ότι, θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι υπήρχε ένα πρόβλημα πολύ χαμηλών το, επιτοκίων και υπερβολικής ε, δαπάνης από πλευράς ε, των κυβερνήσεων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν όχι να, να διασώσουμε τις, τα παλιά μας πιστεύω, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς χειριζόμαστε το θέμα του δημοσίου χρέους στην έκθεση αυτή και έχω κάποιες αμφιβολίες εάν θα πρέπει κανείς να επιμείνει στο επιχείρημα ότι το χρέο του δημοσίου τομέα δεν είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι τομεί όπου έχω αμφιβολίες. Από την άλλη, η πολιτική δεξιά θα πρέπει να δεχτεί ότι η έκρηξη του ιδιωτικού χρέους είναι πρόβλημα και θα πρέπει να ρυθμιστεί. Εάν προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε την ιδεολογία από κάποιες από τις συζητήσεις ε, που έχουν να κάνουν με την κρίση, αν μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό κατά την εξέταση των τροπολογιών, θα έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μία έκθεση η οποία πραγματικά να ενδιαφέρει τους πολίτες και που να μπορέσει να επιφέρει θέμενη αξία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Κομφεράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να κάνω μια σύντομη παρατήρηση για τη μέθοδο εργασίας. Φρονώ ότι είναι χρήσιμο, όπως υπενθύμησαν πολλοί από τους συναδέλφους, να χρησιμοποιήσουμε την εβδομάδα που αποφασίσαμε πριν από λίγο για να συζητήσουμε τις τροπολογίες, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ε, να μην κάνουμε απλή παρουσίαση τροπολογιών, απλώς να υπάρξει μία αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ευρεία συνένεση. Με μία προειδοποίηση εδώ, ε. Η συζήτηση των τροπολογιών ε, είναι κάτι το φυσικό και καθόλου ένομο, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε την εντύπωση ότι θα αλλάξουμε κατεύθυνση. Το μόνο που θα καταφέρουμε αν περάσουμε πολλές τροπολογίες είναι να καταστρέψουμε ένα κείμενο και να το κάνουμε ακατανόητο. Πάντα θεωρώ ότι είναι καλύτερο να υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων παρά να έχουμε ένα συμβιβασμό ο οποίος θα είναι δυσνόητος. Βέβαια καλό θα ήταν να έχουμε όλες τις ίδιες απόψεις. Εγώ προσωπικά προσπαθώ ε, να τηρώ κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν τη συμμερίζονται την άποψή μου και άλλοι, αλλά ίσως είναι πιο αποτελεσματικό. Τώρα, για την έκθεση της Περβάνς, ε, την οποία εξετίμησα ιδιαιτέρως ε, και στις συζητήσεις που κάναμε στο παρελθόν, όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο, αλλά και στο, ε, ως προς την οργανωτική δομή της. Να προσθέσουμε και κάποια πράγματα για τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και τις τελευταίες εβδομάδες, διότι αυτά τα γεγονότα είναι και πολύ σημαντικά, αλλά και πάρα πολύ ευαίσθητα. Και εγώ, όπως πολλοί από εσά, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μας ε, επηρεάσει η κυρίαρχη άποψη ότι ε, το βασικό που μας ενδιαφέρει είναι το χρέος, ε, ο έλεγχος του και η σταθερότητα που θα πρέπει να διασφαλίσουμε για την οικονομία της κάθε χώρας. Δεν θα ήθελα φυσικά βέβαια να πω ότι αυτές τις ε, ε, πτυχές τις θεωρώ ίσονο σημασία, ίσα ίσα είναι πολύ σημαντικές. Αλλά η οικονομική πτυχή για πολύ αυστηρά μέτρα εξυγίανσης δημιουργείται κατά την άποψή μου λαμβάνοντας υπόψη δύο προϋποθέσεις. Την ισοτιμία στις ε, δράσεις εξυγίανσης καθώς επίσης και αξιόπιστες και ρεαλιστικές πολιτικές ανάπτυξης. Εάν δεν τηρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις, το θέμα της εξυγίανσης ουσιαστικά ε, μειώνει την αυστηρότητα και κάνει τους ανθρώπους να είναι αντίθετοι στις πολιτικές εξηγήσεις. Όπως ε, θα γνωρίζουν οι κυβερνήσεις ε, κάθε κράτους μέλους, είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο αυτό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Αν δούμε τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν σε κάθε χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, ε, κυρίως ως προς τις πολιτικές εξηγήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να μην κάνουμε την εξή ε, επίκριση. Από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν ε, υπερισχύει η πειθαρχία και υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποφύγουμε εμεί να διαπράξουμε το ίδιο σφάλμα και το λέω αναφερόμενο σε κυβερνήσει, οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικές πολιτικές ε, αποχρώσεις. Όταν εμεί θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε το κείμενο αυτό στο Κοινοβούλιο, εδώ θα έχουμε εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων Ευρωπαίων εργαζομένων και συνδικάτα όχι μόνο από κάθε χώρα αλλά και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έχουν ήδη προγραμματίσει δημόσιες πρωτοβουλίες που πραγματικά ε, φαίνεται ότι θα έχουν και πάρα πολύ κόσμο και θα είναι πάρα πολύ ισχυρέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν υπάρχει μια προφανής κοινωνική πτωχή και αυτή φυσικά είναι η δυσαρέσκεια που υπάρχει σε κάθε χώρα και υπάρχει κίνδυνος ε, οριστικής ρήξης του κοινωνικού διαλόγου και να απώλειας όλων αυτών των στοιχείων που ήταν κυρίαρχα στην Ευρώπη. Και εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα όχι μόνο για την, Ευρώ... για την Ελλάδα όπου τα μέτρα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά για προφανείς λόγους, αλλά υπάρχουν φαινόμενα ρήξης και σε άλλες χώρες, τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, αυτό το στοιχείο της ισοτιμίας και η πολιτικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι ρητός ε, ε, γραμμένα στις προτάσεις μας. Θα ήθελα να σταθώ και σε αυτό το θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων, το οποίο ανακύπτει από καιρούς καιρών. Πραγματικά, εμένα μου ξεφεύγει ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνεται αυτό. Ε, πάντα ασχολούμαι με εργαζομένους, αλλά ποτέ δεν θα ε, πρότεινα σε έναν εργαζόμενο να επενδύσει τις οικονομίες του στην επιχείρησή του. Γιατί να πρέπει να κινδυνεύει να χάσει και τη δουλειά του και τις οικονομίες του, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ναι, η, η ιδέα της συμμετοχής έχει μια ιδέα λαϊκισμού, αλλά από την άλλη ο εργαζόμενος και ο εργοδότης ε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η εκπροσώπηση αναγνωρίζεται, θα πρέπει να είναι παρόν ο εργαζόμενος για να προασπίζεται τα συμφέροντά του όλα ένα προς ένα, να μην αποκλείουμε κανένα, αλλά από εκεί και πέρα να υπάρχει συμμετοχή ανθρώπων που έχουν ένα πολύ σαφώς καθορισμένο χαρακτήρα στη ζωή μιας επιχείρησης, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνεται πάρα πολλές από τις επιχειρήσεις που απέτυχαν, ε, εάν είχαν συμμετοχή των οργαζομένων αυτή τη στιγμή, θα ήταν σε πολύ δυνότερη κατάσταση από αυτή που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Η Ελίζα Φερέιρα. Muito obrigada. Eu acho que este relatório geral sobre ele parece-me de facto extraordinariamente completo θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο για, αυτό το, για αυτή την έκθεση, η οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετική. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας συγκεκριμένα σημεία. Γιατί όπως είπαν αρκετοί συνάδελφοι, οι Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται σε, σε μια κατάσταση απογοήτευσης. Είναι άνεργοι και απογοητευμένοι από το συνολικό εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτή την έκθεση σαν ε, ένα τρόπο να ξεκινήσουμε πάλι αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα και να θερίνουμε και τα άλλα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δράσουν και να επανατοποθετηθούμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πάλι ελπίδα στον πολίτη για το μέλλον της Ευρώπης. Νομίζω ότι ο παραδοσιακός τρόπος υποβολής τροπολογιών θα διαστρεβλώσει αυτή την έκθεση. Θεωρώ ότι η έκθεση είναι αρκετά αξιόλογη και πολύτιμη. Γι' αυτό θα προτιμούσα να επιλέξουμε τέσσερα θέματα με ξεκάθαρα μηνύματα, τα οποία θα είναι το αποτέλεσμα ε, αυτής της έκθεσης και θα κοινοποιηθούν. Κατά την άποψή μου υπάρχουν τέσσερα θέματα τα οποία θα ήθελα να περιληφθούν σε αυτή την έκθεση ή μάλλον να προέλθουν από αυτή την έκθεση, παρόλο που δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια συνένεση. Το πρώτο θέμα, το οποίο νομίζω, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό, αφορά την ανανέωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να επανατεθούν στην ημερήσια διάταξη. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οικονομικοί, πρωτίστως οικονομικοί στόχοι, είναι πολιτικοί στόχοι, βασίζονται στη δημοκρατία και στην έννοια της ελευθερίας. Αλλά η δημοκρατία και η ελευθερία έχουν βεβαίω και μια οικονομική συνιστόσα, γιατί αν 20% του πληθυσμού μας αποκλείονται και είναι φτωχοί, τότε εξ ορισμού η ελευθερία και η δημοκρατία θα είναι διαφορετική για αυτούς τους πολίτες από ό,τι είναι για τους για την πλειονότητα των υπολείπων πολιτών. Συνεπώς λοιπόν οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να τοποθετούν και πάλι, τοποθετούν στην μερίσια διάταξη. Και αυτό νομίζω αναφέρεται στην ίδια την έκθεση. Το δεύτερο θέμα είναι το εξή. Ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ούτως ώστε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, είναι αναγκαία και η πολιτική αλλά και η οικονομική δημοκρατία και θα πρέπει να διαμορφώσουμε μία εντελώς ε, διαφορετική ημερήσια διάταξη, όχι σαν την παλιά που βασιζόταν μόνο στην εσωτερική αγορά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, αλλά προκειμένου να τεθούν στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής ημερήσιας διάταξης δεν μπορούμε να ορίσουμε τις έννοιες αυτές μόνο πολιτικά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα επιπλέον έργο, μια επιπλέον προσπάθεια για να δούμε πώς η Ευρώπη θα μπορέσει να είναι ελκυστική για επιχειρήσεις να εγκατασταθούν εκεί, γιατί στο πλαίσιο ενός κόσμου θα πρέπει να διασφαλίσουμε οι επενδυτές να προτιμούν να επενδύσουν στην Ευρώπη παρά στην Κίνα ή τη Λατινική Αμερική ή την Αφρική. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο, ένα πιο δομημένο τρόπο σκέψης. Θα πρέπει να σκεφτούμε πιο ξεκάθαρα ποιο είναι το ευρωπαϊκό συμφέρον. Και σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια ε, εξωτερική οικονομική πολιτική. Δεν μιλάω για τον προστατευτισμό, αλλά εννοώ για το πώς μπορούμε να διαφορθώσουμε τις σχέσεις μας με το περιβάλλον παγκοσμιοποίησης προσπίζοντας στα δικά μας συμφέροντα. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις σχέση με τις λεπτομέρειες της χάραξης βιομηχανικής πολιτικής. Υπάρχουν αυτά τα δύο θέματα τα οποία περιλαμβάνονται και στην Ατζέντα 2020 και που είναι νέα σε σχέση με τη συνθήκη Θεσσαλονίκη της Λισαβόνας. Όταν, μιλούμε για, όταν μιλάω για βιομηχανική πολιτική, ε, περιλαμβάνω και τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην έκθεση. Το τρίτο θέμα είναι η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Νομίζω ότι όλες οι θεμελιώδεις ιδέες ε, βρίσκονται εδώ πρέπει να έχουμε μια αποτελεσματική ρύθμιση. Αλλά καθώς με αφορά η οργάνωση των θεσμικών οργάνων που προτείνεται εδώ μετά από τις ε, τελευταίες εμπειρίες θα πρέπει να επαναταθεί επίσης το ζήτημα των ευρωομολόγων, το ζήτημα της ε, φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να αναφερθούν ξεκάθαρα εδώ. Νομίζω ότι η ρύθμιση είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που θα πρέπει να βγαίνει από αυτή την έκθεση. Ένα τέταρτο θέμα, επίσης ουσιαστικό και που αναφέρεται εδώ, ε, στην παράγραφο 59 στο 72 οι προϋποθέσεις για την ε, οικονομική επιβίωση αναφέρεται μεν εδώ, αλλά δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα στην έκθεση και είναι σημαντικό να μιλήσουμε με μια ξεκάθαρη γλώσσα, Οικονομική και Νομισματική Ένωση. με εντελώ διαφορετικού τομεί ανταγωνιστικότητα. Γιατί η ανταγωνιστικότητα εντό τη Ευρώπη ε, ποικίλει. Και χρειαζόμαστε ένα ίσο επίπεδο το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας δεν μας εξασφαλίζει πλέον την πρόοδο. Και ήταν προφανές ευθύς εξ αρχής ότι ορισμένοι τομείς χρειάζονται εσωτερικούς μηχανισμούς αντιστάθμισης που δεν προβλέπονται από τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό, που δεν έχει καταρτιστεί για κάτι τέτοιο από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η απόκληση μεταξύ των διαφόρων τομέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεγαλώσει, οι ανισορροπίες μεγάλωσαν. Και σήμερα θα πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Γιατί το πρόβλημα ε, δεν ε, είναι μόνο το ζήτημα της εθνικής υπερχρέωσης, το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει και βεβαίω θα μπορούσε να σκοτώσει την ε, νομισματική και οικονομική ένωση εκτός αν έχουμε το θάρρος να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό το ερώτημα είναι διαφορετικό από το ζήτημα της ε, απάτης της στατιστικέ. Οι αποδοχέ θα πρέπει να πέσουν, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για να αντανακλούν τα επίπεδα τη παραγωγικότητα, εφόσον δεν έχουμε μηχανισμούς αντιστάθμισης και αυτό θα συνεπιφέρει προβλήματα γιατί αν έχετε μία ένωση όπου το κόστος διαβίωσης ε, είναι περίπου ίδιο σε όλη την Ένωση, θα πρέπει να υπάρχουν παρόμοιες αντίστοιχες αποδοχές. Αλλά αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή και αυτό συνιστά ένα πρόβλημα. Αυτό ήδη αναγνωρίστηκε πριν από 10 χρόνια σε κείμενα σε σχέση με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα παραμένει και, αν, και θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προτάσεις ανάκαμψης που να σχετίζονται με αυτό το θέμα. Αυτά είναι λοιπόν τα τέσσερα θέματα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την έκθεση και να αποτελέσουν τα βασικά του μηνύματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγελ. Εγώ κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ορισμένες φορές δεν έχει νόημα ένα συμβιβασμός αποκυμνωμένος από το νόημά του. Είναι προφανές ότι οι διαφωνίες που υπάρχουν εδώ είναι από ιδεολογική άποψη τόσο μεγάλες που θα μπορούσαμε να οργανώσουμε τη μεγάλη σύγκρουση των πολιτισμών χωρίς να παραχθεί από αυτό καμία απολύτως υπεραξία. Έχω την άποψη ότι αν θέλουμε το έργο αυτό να έχει τελικά μια υπεραξία, θα πρέπει να προσδώσουμε μια πιο ε, σφαιρική ή νέα διάσταση σε αυτό το οποίο συνέβη και βρίσκεται υπό εξέλιξη γιατί η Ευρώπη δεν τοποθετείται ούτε εντελώ δεξιά ούτε αριστερά, απολύτω στην αριστερά. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε ένα κείμενο το οποίο είναι σοσιαλιστικής έμπνευση ή από, να εμπνέεται από μια δεξιά λογική. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα, ότι το κάνει πιο θεμητό στα μάτια εκείνων που περιμένουν από εμά συγκεκριμένα συμπεράσματα. Εγώ... Ε, υπάρχουν πολλοί που λέει ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα μείζωνα θέματα. Μίζωνα θέματα από τα οποία θα υπάρξουν σίγουρα διαφωνίες, όπως για παράδειγμα το δημόσιο χρέος η εξέλιξη του χρέους στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις του. Θα πρέπει να έχουμε συνείδηση του γεγονότος και θλίβομαι για την αριστερά ότι το επίπεδο του χρέους στην Ευρώπη ήδη πριν από την κρίση είχε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα σε εποχές ειρήνης, ιστορικά επίπεδα. Δεν μπορούμε να περάσουμε τη γέφυρα και να πούμε ότι εντάξει καλά ζήσαμε, ας συνεχίσουμε να ξοδεύουμε θα πρέπει να δούμε τι θα καταφέρουμε αν συνεχίζουμε να ξοδεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό στη, στο Νότο το διαπίστωσαν ήδη, αλλά θα το διαπιστώσουμε και στο Βορρά. Εγώ έχω την άποψη ότι δεν υπάρχουν, ε, δεν έχουμε καμία πλέον κανένα περιθώριο ε, δαπάνης, κατανάλωσης και είναι αυτό το θέμα, αυτή η αντιπαράθεση σχέση με την ε, λιτότητα και την ε, μεγέθυνση, όπου κατά την άποψή μου θα πρέπει να τεθεί περισσότερο με όρους ανάγκης της λιτότητας από τη μία και της ανάπτυξης που θα πρέπει, του τρόπου ανάπτυξης που θα πρέπει να απορρεύσει από την πολιτική λιτότητας. Και εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη αυτή η αιμονή της ανάπτυξης, της μεγέθυνσης, μοιάζει με αυτή την αιμονή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ δεν έχω τίποτα κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν είναι όμως σαν να είχαμε ένα εικοστό πρόγραμμα, πρόγραμμα υπέρ των, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, έτσι θα ξεπερούσαμε την κρίση και θα υλοποιούσαμε την πλήρη απασχόληση. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Και νομίζω ότι αυτός δεν είναι ο δεδομένος τόπος για να περάσουμε στο 28ο πρόγραμμα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά μάλλον για να καταλήξουμε σε μια ανάλυση της κατάστασης που μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν μπορούμε, ιδίω στην Ευρώπη, αλλά γι' αυτό μιλούμε, ε, ε, έχω την εντύπωση, δεν μπορούμε στο δυναικές να επινοούμε και πάλι και πάλι νέα μέτρα ανάπτυξης μέσω δημοσίων δαπονών που τελικά δεν χρησιμεύει από το να διατηρεί το σύστημα κοινωνικής ε, ασφάλισης σε, ένα, σε μια συνεχή ανισορροπία. Και βρίσκεται ακριβώς το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης στο επίκεντρο της συζήτησης, γιατί σχετίζεται με τις μας δαπάνες. Το 62% στη δική μου χώρα του κρατικού προπολογισμού ε, ε, σχετίζεται με αυτό. και συνήθως χαρακτηρίζονται ως μη κατανοητές αυτές οι δαπάνες. Ε, τότε θα σταματήσουμε αμέσω ή να θεωρήσουμε ότι στη Νότια Ευρώπη θα γίνουν κάποια θαύματα, γιατί απαιτούμε από την Ελλάδα, από την Πορτογαλία, από την Ισπανία και στους από την Ιταλία και άλλες χώρες μέλη, μία πολιτική λιτότητα που θεωρώ ότι σε άλλα, άλλους τόπους της Ευρώπης λειτουργεί. Στη Λετωνία λειτουργεί κάτι τέτοιο, όσο παράδοξο και να φαίνεται γιατί μπορεί να υπήρξε αποπληθωρισμός μέσω των, ε, των αποδοχών, όπως λέει η συγκήτρια, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια ποσοστά ανάπτυξης. Ίσως αυτό φαίνεται σαν ένα θαύμα. Υπάρχουν λάστιοι οικονομολόγοι που να μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί συνέβη κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά το θαύμα υπάρχει. Και ε, είτε στη Λούρδη είτε στη Φάτιμα είτε οφείλεται σε άλλους παράγοντες, δεν ξέρω. Για μένα ε, θεωρώ ότι μοιάζει να λειτουργεί. Και τα διδάγματα που μπορούμε να αντιλήσουμε από μια τέτοια πολιτική είναι ορατά. Αλλιώς γιατί θα πετύσουμε από όλε αυτέ τι χώρε του Νότου να υποβληθούν σε μέτρα λιτότητα. Σίγουρα αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Εάν δεν περιμένουμε από αυτή την πολιτική λιτότητας μία καμπή, ούτω ώστε επιτέλου να υπάρξει εξυγίανση και ανάκαμψη. Και τέλος, ένα τελευταίο, μια τελευταία παρατήρηση στο θέμα της διακυβέρνηση. Θα μπορούσα να πω ότι θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι, γιατί δεν είμαι 100 χρονών, αλλά κάπου διάβασα και περισσότεροι από εμάς το έκανα επίσης, ότι το 29 ο προπολογισμό των ΗΠΑ ήταν 1% του ΑΕΠ. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να μας εμπνεύσει κάποια διδάγματα, γιατί ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι περίπου 1% του ΑΕΠ. Είναι 1,2 ίσως, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ παραπάνω από το 1. Αυτό που για μένα σημαίνει ότι στο μέτρο που υπάρχουν ε, υπάρχουν πολλές διαφωνίες σε επίπεδο θεσμικών οργάνων στην Ευρώπη όσον αφορά τον αναδειγμένο τρόπο προσέγγισης κατάσταση στο μέτρο που οι αρχές του προϋπολογισμού ή μάλλον η εθνική κυριαρχία σε ζητήματα προπολογισμού στην Ευρώπη έληξε. Στο μέτρο που προσπαθούμε να βρούμε νέες συνταγές που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν ένα καλύτερο κοινοτικό προπολογισμό, ίσως ήρθε η στιγμή να πούμε ότι θα πρέπει να περάσουμε σε μεγαλύτερη ταχύτητα όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και αυτό όχι μόνο για να ισχύσουμε το ένα ή το άλλο θεσμικό όργανο. Μ' αρέσει η παράγραφος 154 περβάς. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Αλλά θεωρώ ότι ίσως ε, θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν περιμέναμε ακόμα έξι μήνες θα μπορούσαμε τότε να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για μια ομόσπονδη δομή με έναν προπολογισμό που ίσως θα μπορούσε να μας χρησιμεύσει και ίσως θα έπρεπε να είναι μία από τις φιλοδοξίες της Επιτροπής να διατυπώσει αυτό το στόχο αρκετά, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Και εγώ θα ήμουν υπέρ αυτών που υποστηρίζουν μία τέτοια προσέγγιση. Κοίταξε Συγγνώμη, εσείς ήσασταν πρώτοι. Η Άννη Ποδηματά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επί του διαδικαστικού θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου με την παράταση κατά μία εβδομάδα που δόθηκε για να υπάρχει επαρκής χρόνος ε, και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουμε σε ένα κοινό ε, συμπέρασμα σε σχέση με την ε, ε, έκθεση της Περβάνς Μπερές. Ταυτοχρόνως όμως ήθελα να επισημάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει το Κοινοβούλιο να εγκρίνει εγκαίρως αυτή την έκθεση πριν να κλείσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές διότι ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στο μέσο της κρίσης, η κρίση εξελίσσεται και μάλιστα μετεξελίσσεται, έχει πολύ μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει αντανακλαστικά ε, και να απευθυνθεί στους Ευρωπαίους πολίτες με μια τολμηρή και περιεκτική έκθεση σε ό,τι αφορά τα αίτια και τις προτάσεις εξόδου από την ε, σημερινή κρίση. Και ε, υπ' αυτό το πρίσμα θεωρώ εξαιρετική την έκθεση της Περβάνς Μπερές... κυρίως ε, γιατί εστιάζει και εμβαθύνει ε, επαρκώς στα αίτια της σημερινής κρίσης, διότι πιστεύω ότι αν δεν είμαστε ακριβείς και ουσιαστικοί στον προσδιορισμό των, ε, των αιτιών και μείνουμε σε μια επιφανειακή ε, ανάλυση ε, των αιτιών που μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση, δεν θα είμαστε στο, ύψος των, στο των περιστάσεων. Ποιο είναι ο βασικός στόχος κατά τη γνώμη αυτής της τη και της δουλειά που γίνεται σε αυτή την Επιτροπή. Ο βασικός στόχος θεωρώ ότι είναι ακριβώς να εμβαθύνουμε ουσιαστικά στους λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε εδώ, ε, με δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι ε, να βγάλουμε εκείνα τα συμπεράσματα ε, και να διατυπώσουμε τις προτάσεις εκείνες που θα περιορίσουν ή θα αποτρέψουν τις πιθανότητες να επαναληφθούν αντίστοιχες κρίσεις στο μέλλον. Αυτός είναι ο ένας στόχος αυτής της έκθεσης και της δουλειάς που γίνεται εδώ. Και ο δεύτερος στόχος Εξίσου σημαντικός είναι να βρούμε τρόπους και να διατυπώσουμε προτάσεις για να αμβλύνουμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης που διανύουμε σήμερα στους πολίτες, στην ποιότητα της ζωής τους, στην εργασία τους, στην ασφάλεια που πρέπει να αισθάνονται για το ε, παρόν και το μέλλον τους. Αυτή, αυτή κατά τη γνώμη μου, ε, είναι, αυτό είναι το βασικό μας διακύβευμα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θέλω να έρθω ε, στην υπόθεση των, των αιτιών για την οποία έγινε μεγάλη συζήτηση και σήμερα εδώ στην ε, Επιτροπή να κάνω τις εξής πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη αυτήν εδώ την Επιτροπή και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για το ελληνικό ζήτημα. Έχουμε επισημάνει κατά επανάληψη τις ελληνικές ευθύνες. Έχουν αποδοθεί οι ελληνικές ευθύνες, οι ευθύνες του Ευρωπαϊκού Νότου γενικότερα. Θα έλεγα μάλιστα ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που ε, πληρώνεται το τίμημα αυτών των ευθυνών. Ταυτοχρόμως όμως νομίζω ότι με βάση ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή το εύρος και η έκταση της κρίσης, εντός αλλά και εκτός ευρωζώνης πλέον, δεν θα ήταν ιδιαίτερα πιστικό για τους πολίτες και δεν θα ήταν και πολύ παραγωγικό για τη δουλειά που κάνουμε να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια της σημερινής κατάστασης μόνο στο ελληνικό ζήτημα, θα έλεγα γενικότερα μόνο στις ευθύνες του Ευρωπαϊκού Νότου. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, ε, το ΑΕΠ της Ελλάδας αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ του Ευρωπαϊκού. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι θα είμαστε στο ύψος των περιστάσεων εάν επικεντρώσουμε την προσοχή μας ως προς το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ε, στις ε, παρατεταμένες δημοσιονομικές εκτροπές από την πλευρά της Ελλάδας και γενικότερα της χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου. Νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα δομικά, σοβαρές αδυναμίες στη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και βεβαίως στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, στο έλλειμμα παγκόσμιας οικονομικής ε, διακυβέρνησης, τη στιγμή που οι αγορές είναι παγκοσμιοποιημένες, είναι ισχυρές, είναι διασυνδεδεμένες. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτονόητα, είναι πέρα από ιδεολογικοπολιτικές διαχωριστικές γραμμές, είναι απλώς ε, επισημάνσεις ε, που είναι σοβαρές και ορατές για όλους μας. Το θέμα, ένα, ένα θέμα λοιπόν είναι γιατί. Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό και περισσότερο σημαντικό ζήτημα είναι που πάμε από εδώ και πέρα. Και επ' αυτού υπάρχουν πολύ ε, ουσιαστικές προτάσεις και στην έκθεση της Περβάνς και πολύ σημαντικά πράγματα λέχθηκαν και από τους συναδέλφους στη διάρκεια της σημερινής συζήτησης. Χρειαζόμαστε μια αυστηρότερη εφαρμογή και μια καλύτερη υποπτία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να έχει αντίρρηση επ' αυτού. Ταυτοχρόνως όμως θέλω να προσθέσω ότι αυτό που δεν χρειαζόμαστε στον τρόπο με το οποίο σχεδιάζουμε το μέλλον είναι νέες διαχωριστικές γραμμές. Ε, οι νότιοι και οι βόρειοι, τα παλιά ε, και τα νέα κράτη-μέλη. Είναι βέβαιο ότι αν υπάρχει ένα συμπέρασμα που βγαίνει από την παρούσα κρίση είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, άρα μεγαλύτερη και περισσότερη συνοχή μεταξύ μας, ασφαλώς καλύτερη εφαρμογή ε, των κοινών κανόνων, αλλά και μια ισορροπία ανάμεσα ε, στους κανόνες που θα μας εξασφαλίσουν όχι μόνο την ορθότερη δημοσιονομική ε, σταθερότητα, την ορθότερη, την καλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή, Χρειαζόμαστε μία ισορροπία ανάμεσα σε κανόνες που θα μας διασφαλίζουν ασφαλώς την δημοσιονομική ε, προσαρμογή, τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά ταυτοχρόνως θα προστατεύουν ε, την απασχόληση και θα διασφαλίζουν τον μέλλον μας προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα τελευταίο σημείο. Γίνεται μεγάλη συζήτηση ε, στην Ευρώπη και παγκοσμίω θα έλεγα, αλλά ε, ιδιαίτερα στην Ευρώπη ε, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, ε, με αφορμή τη γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού, των ασφαλιστικών συστημάτων. Γίνεται συζήτηση στη Γαλλία, γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα, γίνεται συζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να επισημάνω ότι απουσιάζει οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση και πρόταση για την αναχέτηση αυτής της τάσης, της γύρανσης δηλαδή του ευρωπαϊκού πληθυσμού και τη συνεχής, συνεχούς μείωσης του ε, ε, αριθμού των γεννήσεων. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια τεράστια πρόκληση για την Ευρώπη που χρειάζεται άμεσα γενναίες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας περιορίζοντας τις λύσεις που προτείνουμε στην αναμόρφωση των ασφαλιστικών συστημάτων. Είναι, είναι αναγκαίο μέτρο, αλλά δεν θα μας λύσει το πρόβλημα και δεν θα το αντιμετωπίσει στην ρίζα και στην ουσία του. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να θέσουμε ως βασική προτεραιότητα την ε, προστασία και την ενθάρρυνση με ε, γενναία κίνητρα των γεννήσεων στην Ευρώπη, κίνητρα που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εξαιρούνται και το λέω αυτό με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αυτή την περίοδο που θα πρέπει να εξαιρούνται από τα προγράμματα ε, περικοπών και δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως θα έπρεπε αυτή την πρόσθετη εβδομάδα που ε, μας δίδατε τώρα να την εκμεταλλευτούμε. Να σκεφτεί ο καθένας τι μηνύματα θέλει κάθε πολιτική ομάδα να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Διότι μπορεί να συμπεριλάβουμε πράγματα τα οποία αργότερα να θεωρηθούν ιστορικά. Ε, χρήσιμο θα ήταν πέρα από την ανάλυση να καταλήξει το Κοινοβούλιο σε συμφωνία ότι χρειαζόμαστε τελείως ανεξάρτητους ελέγχους των ε, χρηματοοικονομικών αγορών. Θα ήταν χρήσιμο να ενεργήσουμε προληπτικά για να αποφύγουμε τους κινδύνους επίσης σημαντικό για μας αλλά και για τους πολίτες θα ήταν μέτρα της Κομισιόν. Περισσότερη ε, διαφάνεια κατά τη φορολογία, να κλείσουν τα παραθυράκια η φορολογική παράδοση, η ε, παράδειση, να ε, συντονιστούν με έξυπνο τρόπο τα φορολογικά συστήματα, ώστε οι πολιτικοί να μπορούν να τα επηρεάζουν περισσότερο. Εμένα κάπως με ενοχλεί το ότι θα έπρεπε να είχαμε αναλύσει περισσότερο το σκηνικό αυτό των χρεών. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει καλή και κακή χολυστερίνη, έτσι υπάρχει καλό και κακό χρέος. Όταν μια χώρα λάβει ένα χρέος αλλά το χρησιμοποιήσει για να εφαρμόσει και ενωτόμα μέτρα, αυτό είναι θετικό. Επίσης, υπάρχει μία πτυχή που δεν εξηγείται επαρκώς. Μπορεί να είμαι αφελής, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το κοινό μήνυμα. Η οικονομική πολιτική να διδάσκεται περισσότερο στα, στις επαγγελματικές σχολές, στα πανεπιστήμια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι μόνο χρέη των τραπεζών, δεν είναι κάποια φανταστικά προϊόντα που πολλούνται. Ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει καλύτερα περί τίνος πρόκειται. δεν αρκεί το... Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ε, χαμηλά επιτόκια κατά, τον, ε, κατά τις επενδύσεις και ψηλά κατά, τον, ε, κατά τις επενδύσεις. Η νεολαία είναι σημαντική για το μέλλον. Και πάλι έξυπνοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να δημιουργήσουν νέα προτόντα για να, για να παραπλανήσουν του ε, καταναλωτέ. Ο κόσμο θα πρέπει να μπορεί να ε, κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε καλά και κακά ε, χρηματοοικονομικά προϊόντα. Θα πρέπει να είναι πιο σαφείς οι αξίες. Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την παραπάνω αυτήν την εβδομάδα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να σκεφτούμε τι μηνύματα θέλουμε να μεταφέρουμε στους πολίτες, στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έβαλα και το δικό μου όνομα ε, στον κατ κατάλογο των ομιλητών. Ε, ο συντονιστή μας και η συγητή Όλε ήδη είπε πολλά και άλλοι συνάδελφοι είπαν ε, πολλά από αυτά που ήθελα να πω. Γι' αυτό μπορώ να είμαι σύντομο. Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση σαν τεχνικό όρο και την κρίση που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη. Διότι κατά τη γνώμη μου θα είχαμε την ε, ευρωπαϊκή κρίση ακόμα και χωρίς την παγκόσμια κρίση, διότι στην Ευρώπη ουσιαστικά έχουμε πολιτική κρίση. Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμοι στην Ευρώπη και θα πρέπει να ε, εξετάσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Ε, Έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν, αλλά αν λύσουμε τα προβλήματα αυτά και προχωρήσουμε όπως προχωρήσαμε μέχρι τώρα, αυτό δεν θα αρκεί. Υπόθηκε ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα διαμορφώσουμε την Ευρώπη στο μέλλον. Πρόκειται για μια νέα Ευρώπη, πρόκειται για μια νέα βάση για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες στην κατάσταση των κρατών μελών, στην κατάσταση το, της Κομισιόν και όλων των θεσμικών οργάνων. Αυτό θα πρέπει να το εκφράσουμε σαφώς. Είμαστε επιτροπή που μέσα στο επόμενο εξάμηνο ή δωδεκάμηνο θα πρέπει να ε, υποβάλουμε προτάσεις οι οποίες να μπορούν να εφαρμοστούν. Καλό θα είναι λοιπόν να ε, εκπονήσουμε κάποιες θαραλέ προτάσεις, τολμηρές προτάσεις, τι οποίες όμως θεωρούμε σωστές. Υπόθηκε, αναφέρθηκε το θέμα της περισσότερη Ευρώπης. Για τους περισσότερους αυτό δεν είναι νέο μήνυμα, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να το μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα, πόσο μάλλον να το εφαρμόσουμε. Η δεύτερη μου παρατήρηση, την οποία ήδη ανέφεραν ο Πασκάλ και άλλοι, θα πρέπει τα συμπεράσματά μας να είναι εύληπτα και να είναι διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε ο παραλήπτης των μηνύματων αυτών να μπορεί να τα μεταφέρει και αλλού. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό των πιθανών πολλαπλασιαστών. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε απλά αλλά σημαντικά μηνύματα. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι μήπως θα πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω πάνω στη διαμόρφωση των μηνυμάτων αυτών. Υπάρχουν πολλά μηνύματα που λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση, ε, μας λείπουν κάποια πράγματα, ε, κάποια πράγματα δεν εμπίπτουν στην εντολή μας, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη δομή. Είχαμε μια συνάντηση στο Βερολίνο που ήταν παρούσα και η ε, ε, Περβάνς, ε, εκπρόσωπος της ε, Εθνικής Τράπεζας της ε, Αγγλίας είπε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις δομές. Μήπως χρειαζόμαστε πιο απλές δομές. Το θέμα του δικαίου για την αφαιρεγκαιότητα στην Ευρώπη κλπ. Προτάσεις που να ε, ε, αναφέρονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πώς παρουσιαζόμαστε, πώς εκπροσωπείται ε, σε διεθνή φόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι υποχρεώσεις έχει η Επιτροπή. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Έχουμε επίσης προτάσεις που αφορούν τα κράτη-μέλη. Και εδώ τίθεται το ερώτημα μήπως... Εκτός από την έκκληση να συγκυρίσουν τα χρέη τους, Μπορούμε να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα, μήπως ένα, ε, ε, υπάρχει στο Σύνταγμα των χωρών αυτών ένα φρένο για τα ΑΕΗ. Αυτό είναι μια πολύ αυστηρή απέτηση. Άλλωστε καμία κυβέρνηση δεν τολμά να παραβιάσει το Σύνταγμα, τουλάχιστον όχι επανειλημμένα, κάθε χρόνο. Επίσης θα πρέπει να εκφράσουμε σαφώς το γεγονός ότι η κρίση φαίνεται να έχει... Η τεχνική χρηματοοικονομική κρίση, όχι αυτή της Ευρωζώνης, φαίνεται να έχει υποχωρήσει λίγο. Αυτό όμως είναι πολύ προσωρινό πλεονέκτημα. Πριν λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, δημοσίευσε, νομίζω στην Γερμανία μόνο κιόλας, ότι η ανάγκη για απόσβεση ε, επενδυτικών προϊόντων εκτιμάται σε 200 ε, δισεκατομμύρια ε, ευρώ για, τις, για τα επόμενα δύο χρόνια. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε σαφές ότι δεν αρκεί απλά να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει μέχρι τώρα. Και τελευταία παρατήρηση, μου φαίνεται ότι ε, μπορούμε να έχουμε μία ε, βιώσιμη λύση μόνο εάν ε, όλοι ακολουθούμε τους ίδιους κανόνες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι Κινέζοι κλπ. Να κινούμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Άσχετα από τις τις δηλώσεις φιλίας που ακούμε από τους G20. Αυτό είναι ε, προϋπόθεση εκ των ουκ Αν δεν το καταφέρουν αυτό, τότε ανοίγουμε τις πύλες ε, για ε, ρυθμιστική αυθαιρεσία, για πειρασμούς, ώστε ο καθένας να προσπαθεί να κερδίσει μόνο τόσο γίνεται περισσότερα και έτσι σε κανένα δύο χρόνια πάλι θα έχουμε την ίδια κρίση. Υπερβάνω, έχει την τελευταία λέξη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι υπάρχουν και εκπρόσωποι της Επιτροπής. Θέλουν να πάρουν το λόγο. Όχι. Ε, Ενδεχομένω ε, πίστευα θα μπορούσε να ενδιαφερθεί η Γενική Διεύθυνση, αλλά Εν πάση περιπτώσει ε, θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να περάσουν το μήνυμα που θεωρούν σημαντικό. Καταρχήν ευχαριστώ γιατί πιστεύω ότι η εργασία στην οποία μας κάλεσε ο Ατμαρ Κάρας παρατείνοντας κατά κάποιο τρόπο την ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών έχει ήδη ξεκινήσει. Και νομίζω ότι κάναμε μια συμφωνία λέγοντας ότι η παράταση αυτή της υποβολής τροπολογιών για, ως την 22 Ιουνίου δεν είναι για να παραπλασιάσουμε τον αριθμό των τροπολογιών, αλλά αντίθετα για να προσπαθήσουμε να τις μειώσουμε, που θα ήταν παράδοξο, περισσότερος χρόνος για λιγότερες τροπολογίες. Και ελπίζω ότι θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και αυτή η συνάντηση. Βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα μεθοδολογίας. Η δική μου πολιτική δεν είναι, λέω μιλήτρια, μάλλον η διαθεσιμότητά μου είναι απόλυτη. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα μέχρι την 22 Ιουνίου θα καταστήλ, αναστείλω όλες τις δραστηριότητες για να είμαι απολύτως διαθέσιμη. Αλλά το θέμα είναι το πώς θα οργανώσουμε την εργασία μας, γιατί το είπατε ήδη. Ορισμένοι από εμά είναι στις ΗΠΑ και λοιπά την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, στις πολιτικές ομάδες υπάρχουν κάποια πράγματα που ξεκινούν ήδη αυτή τη βδομάδα, αλλά η προσεχής βδομάδα θα αφιερωθεί στην αναζήτηση μιας ισορροπίας εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, ούτως ώστε αν δεν θέλουμε να καταλήξουμε στη μάχη των τροπολογιών που όλοι είπαν ότι δεν επιθυμούν, θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, ή μάλλον να εξοπλίσουμε αυτή την εβδομάδα, επίσης, ούτως ώστε ο καθένας από εμά να αναγνωρίσει σαφώς τα τέσσερα πεντε βασικά σημεία, μίζωνα σημεία. Αυτή τη στιγμή γίνει η σύνοψη της έκθεσης και να υπάρχει και μία αρμονία μεταξύ των θεμάτων αυτών. Το θέμα είναι, ε, θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί, να πρέπει να το κάνω εγώ με τον καθένα χωριστά. Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να γίνουν και τα δύο. Θα προτείνω ένα ή δύο ραντεβού με τους ε, συντονιστές και τους σκιώδεις την εβδομάδα του Στρασβούργου και θα γράψω προς τους συντονιστές δηλώνοντας τη διαθεσιμότητά, του, τη διαθεσιμότητά μου συγγνώμη, για συνεργασία με τις πολιτικές ομάδες. Τώρα, επί της ουσίας. Σήμερα άκουσα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ε, ενισχύσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ε, αναφερθήκατε στην παράγραφο 153. Είμαστε το μόνο θεσμικό όργανο που μπορεί να κάνει μια τέτοια δήλωση. Πολλοί αναλυτές λένε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιβιώσει στην κλίμακα της ε, παγκοσμιοποίησης είναι ε, το 1930 άρθρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε. Ό,τι υπάρχει στο τραπέζι πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πράγματα που είναι βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Ακόμα και η παράγραφος 64 που αναφέρεται στην οικονομική διακυβέρνηση. Γιατί δεν ζητήσουμε να παραιτηθεί μεθαύριο όλοι η ΡΕΝ και να δημιουργήσουμε μια θεσμική κρίση. Αλλά νομίζω ότι προ αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει η εντολή μα. Έχω αυτή την αίσθηση από την αρχή ότι σε αυτή την ε, ε, ότι εκεί μπορούμε να καταλήξουμε. Το ζήτημα που θα παρουσιάσει δυσκολίες είναι ανάλυση των συνθηκών εξόδου από την κρίση. Και αυτό δεν αφορά μία μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά αυτό που θα κάνουμε αύριο. Είναι οι καταθέσεις που θα θέλουν να οι τροπολογίες συγγνώμη, που θέλουν να καταθέσουν οι βουλευτές για το κατά πόσο θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην Κίνα, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αγαπητέ Φραγκενγκόλ, είμαι η τελευταία. Σε σχέση με το θέμα, να αναφέρω το θέμα της ανάπτυξης ε, πληθωριστικά, όχι αναφέρεται μία ή δύο φορές στην έκθεσή μου. Αλλά δεν ξέρω κοινωνίες που να μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς επενδύσεις. Και αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχονται. Σήμερα γίνεται αποκλειστικά λόγος για το χρέος. Και όπως είπε η κυρία Γιακοντσαρή, το χρέος όταν είναι έξυπνο ισοδυναμεί με μια επένδυση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε πού θα πάμε να ψάξουμε τις επενδύσεις μεθαύριο. Προφανώς οι χώρες μέλη εξάντλησαν τις ικανότητες χρέωσής τους. Και δεν άκουσα καμία διαφωνία. Ε, ιδού και από πού προκύπτει το θέμα των ευρωομολόγων. Γιατί μην κάνουμε τα ίδια ασφάλματα όπως οι χώρες μέλη. Να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα σαν μοχλό για να διορθώσουμε τις ανισορροπίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών μελών και να εξοπλίσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι τη παγκοσμιοποίηση. Τώρα, το χρέος. Εγώ παρακολούθησα την εξέλιξη ορισμένων θεμάτων στο Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια. Στην άλλη άκρη της κλίμακας του χρέους έχουμε το θέμα της ε, χρέωσης, της υποχρέωσης των καταναλωτών. Evolving Credit. Ένας ε, ολέθριος μηχανισμός υπερχρέωσης ιδιωτικής. Και δεν τα πουθενά να καταδικάζει κανείς αυτό το μηχανισμό, που πραγματικά είναι μια μηχανή ολέθρου. Γιατί ε, είναι δυνατόν να χρηματοδοθεί ένα τραπεζικό σύστημα από τη μία ε, θεωρούν όλοι. Από την άλλη λένε ότι το δημόσιο χρέος είναι το μεγαλύτερο δεινό που μπορεί να υπάρξει. Ο κ. Όλε Σμιτ αναφέρθηκε στον ιδεολογικό χαρακτήρα, στην ιδεολογική φύση αυτών των επιχειρημάτων και νομίζω ότι εδώ ανακύπτουν οι δυσκολίες. Το πνεύμα της παρέμβασης της Πασκάλ, του Σέργιο Κοφεράτη, του Ότμαρ Κάρας μας επιτρέπει ίσως συλλογικά να κινηθούμε λίγο πιο έξυπνα. Ιδού λοιπόν δύο παρατηρήσεις γενική φύσεως που ήθελα να κάνω τώρα. Αν με αφήνετε δύο λεπτά θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένου. Φοβούμαι ότι ίσως θα μακρηγορήσω. Εγώ είμαι δεδεθμένη να το κάνω. Έχω κάποια πράγματα να κάνω ήδη απάντηση προς τον κάθε ένα βουλευτή. Αλλά φοβάμαι ότι ίσως αυτό το στάδιο θα είναι κάπως κουραστικό ίσως τηλεγραφικά, για να καταλάβουν οι μεν και οι δε πόσο προσεκτικά άκουσα τα λόγια τους. Κυρία Πετικάινεν δεν είναι εδώ. Άρα τα πράγματα θα είμαι ακόμα πιο γρήγορη. Αυτά που είπε για την Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν αλλάζει τα θεμελιώδη ζητήματα που τίθενται και δεν μπορώ παρά να με αυτή την προσέγγιση και που ανταποκρίνεται σε αυτό που είπε η κυρία Ποδηματά. Η ελληνική κρίση δεν συνέβη επειδή έκανε βλακίες η Goldman Sachs, αλλά επειδή δεν υπάρχει πιλότος στο πιδάλιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, θα μπορούσα να σας παραπέμψω σε κάποιες ε, παραγράφους σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε σχέση με την ε, υποστήριξη των ε, τραπεζών στην παράγραφο 182 και για τη συμμετοχή των εργαζομένων επίσης θα μπορούσα να σας παραπέμψω σε κάποια παράγραφο. Τώρα, κύριε Ντε Νομίζω ότι μοιραζόμαστε πολλά πράγματα όσον αφορά την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Νομίζω ότι υπονομεύεται γιατί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν καλά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στα οποία προσβλέπουν οι πολίτες. Και νομίζω ότι για να συμφιλώσουμε τα πράγματα, το ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι αναμφίβολα ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε. Τώρα, όταν η κυρία Αλβαρέζ επιμένει στο διάσταση της ανάπτυξης του συμφώνου, αυτό είναι ένα από τα σημεία επί των οποίων θα έχουμε δύσκολες συζητήσεις, θα έλεγα, αλλά νομίζω που θα πρέπει να τις κάνουμε. Ο κύριος Τόμασμάν είναι ακόμα εδώ. Άρα θα του το πω, γιατί θα μας επιτρέψει αυτό να ξαναμπούμε σε αυτή που θα είναι το δύσκολο σημείο. Πιστεύω εγώ ότι το να ζει κανείς σε κοινωνία σημαίνει να σέβεται τους κανόνες. Στη Γαλλία θεμελιώδες δικαίωμα ε, είναι ότι η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Αυτό μας επιτρέπει να ζούμε στην κοινωνία. Τώρα, όσον αφορά τον κατασταλτικό ή καταπιστικό χαρακτήρα του συμφώνου, είναι αλήθεια. Αλλά το σύμφωνο δεν αρκεί για να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Αυτό που όλοι λέμε είναι ότι ακριβώς αποσέζει αυτή η προστιθέμενη αξία. Και νομίζω ότι από την έννοια αυτή θα πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε την, ε, ευρωπαϊκή, την ε, μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής και ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και μένα με ανησυχούν οι εργασίες της ομάδας Βαν Ρομπόι που συστάθηκε σε αντάλλαγμα του πακέτου για την Ελλάδα και φοβάμαι ότι θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του, του χαρακτήρα δημοσιονομικής, ε, της πτυχής δημοσιονομικής πειθαρχία του συμφώνου με τον κίνδυνο ότι θα αυξηθεί αυτό το στοιχείο, θα ενισχυθεί αυτό το στοιχείο και τα άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν δεν θα συζητηθούν και θα υπάρξει άρνηση να συζητηθούν τα υπόλοιπα στοιχεία. Και αν συμβεί αυτό δεν θα έχουμε κάνει απολύτως καμία πρόοδο και ίσως αύριο μία ή άλλη χώρα θα βρεθεί μόνη της σε μία κρίση και θα ονειρεύεται ε, σε μια λειτουργία της κοινότητας, αλλά τα πράγματα τότε δεν θα λειτουργούν. Ναι, εντάξει για την πειθαρχία, αλλά μην ξεκινήσουμε από αυτό. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε δημοσιονομική πειθαρχία. Θα επανέλθουμε, αλλά αν ξεκινήσουμε από αυτό θα σκοτώσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία της συζήτησης. Τώρα, σαν αφορά τι παρατηρήσει Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, χαίρομαι που η κυρία προσπίστε τι απόψει. Δεν είχα την άποψη ότι θα τον αφιβόλω το έργο της Επιτροπής. Ε, οι ανακοινώσει αυτέ εκ των υστέρων ήταν πολύ καλέ, αλλά από τη στιγμή που χρειάστηκε να υπάρξει υποστήριξη εκ μέρου των χωρών μελών, οι προποθέσει δεν ορίστηκαν και οι νόμοι που είχε ψηφίσει το Κοινοβούλιο δεν ε, τηρήθηκαν. Ε, όλα αυτά για τα stock options για τους φορολογικούς παραδείσους. Ίσως το κεφάλι της Κομισιόν είχε τις καλύτερες ιδέες του κόσμου, αλλά δεν εμπόδισε τη στιγμή που συστάθηκε το πρόγραμμα υποστήριξης ε, δεν ε, υπήρξε κάποια κίνηση εκ μέρους της Επιτροπής. Κύριε Όλε Σμιτ, συμφωνώ μαζί σας για να πούμε ότι θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, αλλά όχι οποιαδήποτε Ευρώπη. Και όταν λέτε ότι έχουμε ανάγκη την υποστήριξη του κοινού, είναι ακριβώ αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο που αν τους πούμε, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, αν τους πούμε μετά από αυτή την κρίση το μοντέλο το οποίο λειτουργούσε μέχρι τώρα είναι το καλύτερο δυνατό μοντέλο, είναι το καλό μοντέλο, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν υπάρξει μια επάνωδος σε εθνικισμούς και είναι αυτό το οποίο φοβάστε εσείς. Γιατί οι πολίτες ε, δεν έχουν ε, ε, εμπιστοσύνη σε ένα μοντέλο το οποίο έχει εκτροχιαστεί και διαπιστώνουμε όλοι ότι έχει εκτροχιαστεί. Εάν πούμε ότι αυτό το μοντέλο είναι το καλύτερο και συμφωνούμε όλοι για την ανάγκη καταπολέμηση των εθνικισμών, θα καταλήξουμε σε εθνικισμούς. Αυτό που είπατε τώρα για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ένα θέμα το οποίο έχω κατά νου και καλό τον πρόεδρο να το εξετάσει. Έχω το ζήτημα αυτό στο κεφάλι μου εδώ και πολύ καιρό. Και αυτή τη στιγμή συζητούμε για την συνέχιση των εργασιών μου. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι σημαντικό το ζήτημα της σύσταση Εξεταστικής επιτροπή. Κάποια στιγμή το αναφέραν, τα χάθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστασε, ε, συνέστησε συγγνώμη, μία δομή εξέτασης των γεγονότων στην περίπτωση Golden Sachs. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη με μία προσέγγιση εξεταστικής επιτροπής στην Ελλάδα δεν θεωρώ ε, θεωρώ ότι ίσως είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα έπρεπε να διερευνήσουμε περισσότερο αν θέλουμε να παρατείνουμε τις εργασίες μας. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε με το πνεύμα και τα μέσα μιας ουσιαστικής, μια αληθινής εξεταστικής επιτροπής. Μια αντίφαση είναι, θεωρώ, όταν καταλήγεται στο μήνυμά σα αγαπητέ συνάδελφε, λέγεται το καλύτερο είναι το δικό μας μήνυμα και εγώ θέλω να υπάρξει μια συνένεση. Το καλύτερο δηλαδή μας λέτε είναι το δικό σας μήνυμα. Όχι, το καλύτερο είναι μια συλλογική συζήτηση από την οποία να προέλθει ένα μήνυμα στο οποίο να μπορούν να αναγνωριστούν οι περισσότεροι εδώ πέρα. Τώρα για το Πασκάλ. Εγώ είμαι πρόθυμη να κάνω τα πάντα, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Μου, ζητάν, μου ζήτησαν να γράψω ένα ψήφισμα. Αυτό έκανα. Υπάρχουν ορισμένοι σε αυτό το σώμα αναφέρομαι εδώ στον πρόεδρο ότι έχουμε μια ανάγκη να οργανώσουμε την ε, επικοινωνία γύρω από αυτό το ψήφισμα ούτω ώστε να το, κάνουμε εύληπτο. Όσον αφορά την ε, έκθεση, στις τροπολογίες που θα υποβάλω, και θα το κάνω σεβόμενοι τα δεδομένα, αλλά κάνοντας και μια ανάλυση, γιατί έτσι λειτουργώ θα υπάρξουν και συμπληρωματικέ τροπολογίες από την δική μου πλευρά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό παρουσιάζει καμία δυσκολία. Δηλαδή, επειδή με ρωτήσετε αν θα ενημερώσω την έκθεσή μου με τα νέα στοιχεία των τελευταίων εξελίξεων, η απάντηση είναι ναι, θα το κάνω. Τώρα, τα 5-6 σημεία κλειδί όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Η υποχρεώσει διακαθήκοντα ήταν το ε, πνεύμα του άρθρου 173 που θα πρέπει βεβαίω να αναπτύξουμε αλλά στο πλαίσιο της δικής μας συνένεσης εδώ ισχύει. Ναι, και δεν ε, το αναφέρω. Ευχαριστώ που μου τονίζετε τα σημαντικά στοιχεία. Πράγματι συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο. Τώρα η εναλλακτική, η αντιπαράθεση μάλλον, λιτότητα, ανάπτυξη. Αναφέρθηκα σε αυτό και νομίζω ότι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο έξυπνοι για να πετύχουμε κάτι. Τώρα για την Κέι Σουίνμπορν. Είναι διασκεδαστικό γιατί θα ήθελα να της ομολογήσω κάτι. Η ιδέα ότι η κινητικότητα αφορά μόνο τους πλούσιους, mm, μόνο τους στοχούς, αυτή είναι μια ιδέα που δανείστηκα από την Goldman Sachs. Η κυρία Σουίνμπορν αναφέρθηκε στην ανάλυση περιβαλλοντικής διάστασης της κρίσης και τη διασύνδεση με το μοντέλο ανάπτυξης που ήταν το δικό μας. Συμφωνώ μαζί της. Όσον αφορά το δημόσιο νομίζω ότι ήδη απάντησα. Τώρα, για το Σέρτζιο Κονφεράτη. Πολλά από τα σημεία που θέσατε για το θέμα της ισότητας όσον αφορά την εξυγίανση και για μια αξιόπιστη πολιτική ανάπτυξη, δηλαδή το να προσφέρουμε στους ανθρώπους μια προοπτική για το μέλλον. Αυτό, ε, αυτή είναι μια από τις προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση. Και ελπίζω ότι θα μπορέσει να μας κομίσει μια ελπίδα, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Τώρα όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζόμενων. Εγώ είμαι απολύτως σύμφωνη με εσάς όχι μόνο για τους λόγους που αναφέρατε, δηλαδή αυτή τη στιγμή ε, χρεοκοπήσει επιχείρηση, τι θα γίνει με τη συμμετοχή των εργαζομένων ή τι κάνει εργαζόμενος όταν η μετοχή που έχει στην επιχείρηση ε, ανεβαίνει στο χρηματιστήριο σημαντικά και θα έχει την όρεξη βεβαίως να την πωλήσει. Και συνεπώς θα χαθεί ο έλεγχος του κεφαλαίου σε αυτή, στη δομή αυτή. Νομίζω ότι η ιδέα που θα πρέπει να αναπτύξουμε αντίθετα όσον αφορά εναλλακτικέ τύπους ε, εταιρική διακυβέρνησης όπου οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν, θα είναι συγκάτοχοι του κεφαλαιακού δυναμικού της επιχείρησης. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Ε, Λίζα, ε, δεν έχω πρόβλημα με τα όσα είπες για τέσσερα βασικά θέματα. Συγκεκριμένα για το διακύβευμα γύρω από το μοντέλο της Ευρώπης ότι θα πρέπει να είναι ελκυστικό για επενδύσεις. Όσον αφορά τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας, είναι αντικείμενο της παραγράφου 157 αλλά ήδη η ιδέα υπάρχει και θα χαιρόμουν να μπορέσουμε να μάθουμε σε αυτό το σημείο. Ε, για τον κύριο Έγγελ ε, έχει φύγει. Το απάντησα όμως ε, ως προς το τμήμα που μας συνδέει. Σε άλλα πράγματα θα ήμουν πιο κριτική γιατί νομίζω ότι στη Λετωνία άλλωστε είχαμε πάει μαζί και είδαμε μια χώρα που δεν έχει να ζήσει. Δεν είναι μια χώρα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Τώρα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επαγρυπνήσει ούτε ώστε να παραμείνει ένας χώρος καινοτομιών. Ο ιστός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ο ενδεδειγμένος τόπος για να γίνει κάτι τέτοιο. Στην κυρία Ποδηματά νομίζω απάντησα Συγκεκριμένα στο θέμα της γύρανσης του πολιτισμού θα πρέπει να πούμε ότι η αναγνώριση αυτής της πρόκλησης αναφέρεται στην παράγραφο 24, αλλά όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτής της γύρανσης ασφαλώς υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να αναπτύξουμε. Γιατί, τη Λίζα Κοντσάρη, για το θέμα της εκπαίδευσης σε χρηματοπιστωτικά θέματα. Νομίζω ότι θα κουράσουμε τους πολίτες ε, ε, εκπαιδεύοντάς τους, ενώ δεν μπορούμε ποτέ να εκπαιδεύσουμε τους ε, μεγάλους τραπεζίτες που κάνουν τις ακάλυπτες πωλήσει ε, option, τις με συναλλαγές. Οι παρατηρήσεις σας με παραπέμπουν σε μια συζήτηση που είχα πριν από μερικά χρόνια με τον συνάδελφο Ρόμπερτ Γκέμπελς που όταν μας ασκούσαν κριτική κάποιοι για τα συνταξιοδοτικά ταμεία όλοι λέγαμε ότι είμαστε συνένοχοι αυτής της στρατηγικής γιατί θέλουμε να έχουμε τα πιο υψηλά επιτόκια. Αλλά νομίζω ότι η δική σας έκκληση εν σχέση με την αξία του χρήματος και την ηθική αξία είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Αγαπητέ Πρόεδρε, για την ε, πολιτική διάσταση και το γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι που μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτή την Επιτροπή και να το προβάλλουμε σαν μήνυμα. Εκεί όπου θα έχουμε πιο δύσκολες συζητήσεις, πιο τεταμένες συζητήσεις, είναι για τις προϋποθέσεις εξυγίανσης και, το, και την ισορροπία, εξυγίανση και δυνατότητα δημιουργίας ευρωπαϊκής ε, προσθέμενης αξίας. Ευχαριστώ σε όλους επαναλαμβάνω τη διάθεσή μου να συνεργαστώ μαζί σας. Ευχαριστούμε, Περβάν. Στις 3 θα ξαναβρεθούμε.